Sie haben hoffentlich einen guten... Λοιπόν, ελπίζω να είχατε καλές καλοκαιρινές διακοπές όλοι και να γυρίσατε με όρεξη για δουλειά, να γεμίσατε τις μπαταρίες σας. Οπότε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και με τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα έχετε την ημερήσια διάταξη. Ζητήθηκε μία αλλαγή Κάποιο ζήτησε σήμερα το πρωί να προσθεθεί ένα σημείο. Αλλά κάποιοι δεν μπορούν. Θα δούμε. Έχετε κάποιε επιθυμίες για αλλαγή τη ημερησία διάταξη, Όχι. Λοιπόν, εγκρίνεται όσο έχει η ημερησία διάταξη. Σημείο 2 είναι η έγκριση των πρακτικών της 30 η Ιουνίου. Όπω πάντα, αν μέχρι τέλους της συνεδρίασης δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα θεωρηθεί ότι κυρώνονται αυτά τα πρακτικά. Και μετά περνάμε στο σημείο 3. Ανακοινώσεις. Σήμερα αφενός θα έχουμε μια αντιπροσωπεία από την Ινδονησία ανάμεσά μας. Δεν ξέρω αν έχει ήδη φτάσει αυτή η αντιπροσωπεία και μια αντιπροσωπή από την Κένια με τους αρμόδιους υπουργούς εμπορίου που τους καλωσορίζουμε θερμά και καλώς ήρθατε. Έχουμε επίσης ως ήθιστε μία φορά αναέτος μία συνάντηση με τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκινούμε εκπροσώπους των κοινοβουλίων, του Κοινοβουλίου. Στις 6 Σεπτεμβρίου Τρίτη θα γίνει αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι είναι θερμά ε, προσκεκλημένοι. Τους προσκαλούμε θερμά σε αυτή την εκδήλωση. Από τις 18 22 Ιουλίου είχαμε μια αντιπροσωπεία για την UNCTAD που πήγε στο Ναϊρόμπι. Η αντιπροσωπεία αυτή ήταν πολύ επιτυχής. Είχαμε πολλές διμερείς συναντήσεις αλλά και για την εντολή και τη διαμόρφωσή της ε, για την, να επηρεάσουμε τα πράγματα και πολλές συζητήσεις που έγιναν για το μέλλον όσον αφορά την, ε, το ευρωπαϊκό πρότυπο και τις ε, σχετικές δράσεις. Θα δοθεί μια έκθεση στην επόμενη συνεδρίαση και θα τα συζητήσουμε. Ο Αυστραλός Υπουργός Εξωτερικών την επόμενη Πέμπτη θα είναι παρόν στις Βρυξέλλες και θα έχουμε και μια κοινή τότε συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ Επιτροπή Εξωτερικών το πρωί στις 8 Σεπτεμβρίου πρωινή συνεδρίαση. Από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών η αντιπροσωπή από την Ινδονησία μέλη του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας παρίστανται ήδη Καλωσορίζω θερμά τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από την Ινδονησία που θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας και είναι πολύ καλό αυτό διότι η Ινδονησία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια εταιρική συμφωνία που έχει συναυθεί τον Αύγουστο ήδη ώστε η Ινδονησία με αυτόν τον τρόπο να είναι η πρώτη χώρα η πρώτη χώρα που όσον αφορά αυτές τις άδειες, ε, την ε, άδεια ε, license, την παραλαμβάνει ώστε σε σχέση με τις εξαγωγές να γίνονται υποπιστοποιημένες προϋποθέσεις και όρους. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν τους συναδέλφους από την Ινδονησία. Η Ρωσία τώρα και εμείς ενώπιον του ΠΟΕ έχουμε κάποιες κάποια θέματα που εκκρεμούν. Ένα θέμα είχε ολοκληρωθεί και η Ρωσία έχασε, ήταν μια προσφυγή, ένα επίδικο θέμα για δασμούς εισαγωγών και για τα ε, όσα απαιτούνται για τις εισαγωγές αυτές αυτών των ε, αντικειμένων. Είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο παραβίασαν τους όρους του ΠΟΕ Υπάρχουν θέματα λοιπόν που εκκρεμούν. Είναι η πρώτη φορά όμως που η Ρωσία από τον ΠΟΕ πράγματι ε, ε, ε, έτυχε επίπληξης και καταδικάστηκε. Τέλος ανακοινώσεων, σε αυτή τη συνεδρίαση μπορείτε, μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από το διαδίκτυο. Πάρα πολλοί συνδέονται με το διαδίκτυο και παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας τους ε, χαιρετίζω από τη Λισαβόνα, το Ταλίν, την Βουδαπέστη και όλες τις άλλες πρωτεύουσες και όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Τους χαιρετίζουμε όλους. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ανακοινώσεις Προέδρου. Και περνάμε τώρα, θα περνούσαμε ουσιαστικά τώρα, στους κανόνες εισαγωγές για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα από τη Λευκορωσία. Ο κύριος Τάκουλα, εισηγητής, δεν μπορεί να παραστεί αλλά θα εκπροσωπηθεί και δίνω τον λόγο ακριβώς στον συνάδελφο που θα τον εκπροσωπήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ε, δώσω τα στοιχεία που μόλις παρέλαβα, μια που ο Χάνιου δεν μπορεί να έρθει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σύντομα συζητήσαμε και πριν από τις θερινές διακοπές, η έκθεση αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα. Κάποιοι από εσά θεωρήσατε ότι είναι και πολιτικά όμω σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διαγραφούν οι αυτόνομες δασμολογικέ ποσοστώσει κλωστεφαλουργικών ε, ε, προϊόντων και ένδυση από τη Λευκορωσία. Είναι μια χειρονομία θετική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει ότι υπάρχουν σχέσεις εμπορικέ ανάμεσα σε εμά και τη Λευκορωσία. Είναι σημαντικό τρόπο να στηρίξουμε και τον εξυγχρονισμό τη ε, οικονομία τη Λευκορωσίας και υπογραμμίζει ότι έτσι κι αλλιώς δεν ε, έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δείχνει ότι αν υπάρχουν παραβιάσεις υπάρχουν και συνέπειες. Ε, δεν θέλουμε λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά, εφόσον θέλουμε την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ο Χάν υπογραμμίζει ότι σημειώνει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει κάποιοι συνάδελφοι κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό ε, συνέταξε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 17η Σεπτεμβρίου πια. Με τον τρόπο αυτό λέει ότι θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και των κοινοβουλευτικών εκλογών που θα λάβουν χώρα στη Λευκορωσία στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι συνέπειες πάντως ε, στην εισαγωγή κλωστεφατουργικών και ένδυσης από τη Λευκορωσία θα είναι η διαγραφή από το βασικό κανονισμό όλων των διατάξεων που αφορούν τις ποσοστώσεις σχετικά με το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης. Οι ποσοστώσεις αυτές ισχύουν για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλωστιφαντουργικά, τα οποία μετατρέπονται στη Λευκορωσία και επανεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσοστώσεις αυτές σχετικά με το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης δεν ισχύουν για την ε, Λευκορωσία και έτσι αυτό το λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, οι οποίες επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά δεν το είχε λάβει απόψη, επαναφέρουν την κατάσταση όπως πρέπει. Οι τροπολογίες αυτές στο σχέδιο έκθεσης έχουν άτυπα συζητηθεί ήδη με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται ότι εγκρίνονται. Οπότε έτσι μπορεί η νομοθετική αυτή διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση να περάσει. Ο Χάνου προσβλέπει στα σχόλιά σας, τα οποία ε, φυσικά και θα εξετάσει ενδελεχώς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδης εισηγητής, παρακαλώ, στη συνέχεια έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, επεσήμανε η συνάδελφος, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική ε, και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Το αίτημα του εισηγητή με το οποίο συμφωνώ, δηλαδή ε, να υποβληθούν, ε, ε, να περιμένουμε μάλλον τις τροπολογίες ε, μέχρι τα αποτελέσματα των εκλογών στη Λευκορωσία για να δούμε πόσο μεγάλη σχέση έχει ο εμπορικός τομέας με τα πολιτικά στοιχεία της χώρας. Τα βήματα που έκανε η Λευκορωσία, την αποφυλάξη κάποιων πολιτικών κρατουμένων είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά επίσης είχαμε και συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Εράσμους, εξυγχρονισμό και κυρίως ε, προγράμματα ανταλλαγών ε, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τεχνικής και εμπορικής πλευράς έχει αξιολογήσει τι συνέπειες υπάρχουν και τι αντίκτυπος υπάρχει ε, ε για αυτές τις ανταλλαγές. Επομένως, είναι πιο σημαντικό να υπάρχουν εγγυήσεις προς την Ευρώπη ε, και στο σύστημα της κλωσταφαντουργίας μας ότι δεν θα υπάρξει κάποια ζημία ή ε, κίνδυνος ζημίας ε, λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία. Η ε κινδυνος ζημιας λογω της καταστασης στη λευκορωσια η πολιτικη μου ομάδα λοιπόν θα υποστηρίξει την πρόταση και όσον αφορά την κατάργηση των ε, δασμολογικών ποσοστάσεων αλλά και για την ε, σημασία που έχει σε πολιτικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Καρολίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι πρόκειται για σημαντική απόφαση εδώ και ότι τα δημοκρατικά αυτά θέματα για τη Λευκορωσία πρέπει να, είναι, να αναγνωριστούν και θα πρέπει η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας να δούμε ότι συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί. Η κατάργηση των ποσοστώσεων για τα κλωστοϊφαντουργικά για τη Λευκορωσία θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα και οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας θα πρέπει περαιτέρω έτσι να βελτιωθούν. Οι επιπτώσεις σε σχέση με την κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων είναι μικρές, αλλά είναι ένα θετικό μήνυμα που στέλνουμε προς τη δημοκρατία της Λευκορωσίας και συμφωνώ έτσι με τον εισηγητή καταδείχθηκε ότι η απομόνωση δεν βοηθά με κανένα τρόπο για την ανάπτυξη της Λευκορωσίας. Θα ήταν λοιπόν κάτι να δείξουμε και να δούμε τι συμβαίνει στην Λευκορωσία. Είναι σκόπιμο λοιπόν για να αναμείνουμε τις εκλογές, κοινοβουλευτικές εκλογές της 11 Σεπτεμβρίου και σε σχέση και με την Αυστρία με τα θέματα της, ε, ε, των μη διακρίσεων και στην, ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ανώτερη Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά τις εκλογές θα έχουμε επαφή και θα ανταλλάξουμε απόψεις για να αποφασίσουμε αν είναι δυνατόν αυτή η ποσόστοση να καταργηθεί. Είναι σημαντικό σε αυτή την οδό προσέγγισης της Λευκορωσίας προς τα κράτη δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμουμε. Αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε και να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές ε, σε σχέση για παράδειγμα με την κατάργηση της ποσόστοσης αυτής. Ευχαριστούμε. Ο κ. Κάμπε δεν παρίσταται. Α, παρακαλώ. Θα γίνω David Campbell ε, σήμερα το πρωί. Καλημέρα σε όλους, ορίσαμε όλοι. Ε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου και των όσων συμβαίνουν στα υπόλοιπα ε, κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ε, και πρέπει να στείλουμε και ένα στεναρό πολιτικό μήνυμα, ότι αν θέλουμε να χαλαρώσουμε τα μέτρα καταπίεσης και καταστολής, τότε εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Ε, βεβαίως η Λευκορωσία πόρο απέχει από ε, μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη δέσμευση μαζί του καθώς προοδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να είναι βέβαια αργή η πρόοδος και να υπάρχουν και πολλές ε, ε, ε αποτυχίες, αλλά προχωράει. Συμφωνώ με κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις επικείμενες εκλογές στη Λευκορωσία. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών πριν χαλαρώσουμε τις ποσοστώσεις. Ε, μήπως ε, θα στείλουμε και παρατηρητές στις εκλογές. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε Υπάρχουν ήδη 480 διαπιστευμένοι παρατηρητές, αλλά οι 420 είναι από, τις, ε, από την κοινοπολιτεία. Επομένως, ε, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση να το εξετάσει και η Επιτροπή. Ευχαριστούμε. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εύχομαι σε όλους μια επιτυχή εκκίνηση στο υπόλοιπο του 2016. Μπορώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και εμείς ως ε, Νοτική Αριστερά υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση του εισηγητή. Ίσως μια πρόσθετη παρατήρηση πολιτικής, ε, πολιτικού χαρακτήρα σε σχέση με την προετοιμασία της Λέσχης των 20 για την Σύνοδο Κορυφής και μεταξύ άλλων θα πρόκειται και για την τοποθέτηση των της ομάδας των 20 για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού συστήματος και των εμπορικών σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό σε σχέση με τη Λευκορωσία. Διότι είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΠΟΕ και θέματα για τα οποία πώς αντιμετωπίζονται χώρες μη μέλη του ΠΟΕ πώς ε, μπορεί να υπάρξουν σχέσεις με τέτοιες χώρες και να προχωρήσουν, αυτό συσχετίζεται πολύ με την κατάργηση τέτοιου είδους ε, περιορισμών και ε, σε σχέση με την ανταλλαγή εμπορευμάτων και αγαθών. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση του εισηγητή και να δώσουμε την έγκρισή μας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Good morning everybody. Καλημέρα. Είμαι στη Γενική Διεύθυνση Trade στην ε, μονάδα που ασχολείται με την Λευκορωσία. Θα ξεκινήσω με μία μικρή ανακοίνωση γιατί είμαι υπεύθυνη και για τη Ρωσία και είπατε ε, ότι κέρδισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, περίπτωση για τους δασμούς με τη Ρωσία. Αλλά υπήρχε και μια δεύτερη περίπτωση. Έχουμε δύο, δεν είναι μόνο μία στον ΠΟΕ, δηλαδή κατά της Ρωσίας. Για τη Λευκορωσία τώρα, ήμουν ήδη εδώ τον Ιούλιο όταν συζητήσαμε επί της ουσίας, οπότε δεν θα επαναλάβω όλα τα σημεία συμφωνούμε με την κατάργηση και τα όσα ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ε, ε, παθητική τελειοποίηση. Όσον αφορά τώρα τις επερχόμενες εκλογές στη Λευκορωσία, ε, φυσικά και εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση και όταν θα έχουμε περισσότερα φυσικά και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες. Το δεύτερο. Για το γεγονός ότι δεν είναι μέλος του ΠΟΕ η Λευκορωσία. Μπορούμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις με χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ, Για παράδειγμα, θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν, που ούτε και αυτό είναι μέλος. Αλλά η Λευκορωσία θέλει και θα επιταχυνθεί η διαδικασία για τη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε, η κυρία Ρής. Όχι. Όλα σαφή λοιπόν έχουν αποσαφινιστεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 19η Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 19 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Στη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε για αυτές τις τροπολογίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα σε τρία σημεία τα οποία ανήκουν από κοινού σε ένα κοινό πλαίσιο. Το πρώτο είναι η συζήτηση για έξι κατεντολήν κατεξουσιοδότηση πράξης κατεξουσιοδότηση κανονισμούς που αφορούν έξι χώρες που εξαιρούνται πλέον από τις ρυθμίσεις επειδή με αυτές τις χώρες, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις βρισκόμαστε υπό, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις υπό εξέλιξη και επιπλέον και με την Ανατολική Αφρική συναρτάται αυτό και σε αυτό το σημείο χαίρομαι ότι ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου της Κένιας είναι παρόν και θα του δώσω τον λόγο να παρέμβει και υπάρχουν και υπάρχει και το θέμα του ότι η Γκάνα την προσωρινή συμφωνία για την Δυτική Αφρική την έχει προσυπογράψει. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε ε, αλληλοδιάδοχα στη συνέχεια. Ξεκινάμε με τις έξι κατεξουσιοδότηση πράξεις που με βάση τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ όσον αφορά τις ε, διαδικασίες πρόσβασης στις αγορές ε, εξαιρούνται Μποτσουάνα, Κένια, Γκάνα, Ναμίμπια και ε, την θα λάβει τον λόγο αρμόδιος εισηγητής και μετά οι συνάδελφοι θα παρέμβουν εφόσον επιθυμούν. Η απόφαση για τη διαδικασία αυτή θα ληφθεί στη συνάντηση των συντονιστών που θα διεξαχθεί στη συνέχεια. Είναι σαφή. Θα ακούσουμε πρώτα τη γνωμοδότηση του αρμόδιου εισηγητή και θα έχουν όλη τη δυνατότητα έτσι να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν. Και θα αποφασίσουν οι συντονιστές στη συνέχεια τι θα γίνει. Είναι μια συμπυκνωμένη, ας το πω έτσι, διαδικασία αυτή. Προτού ξεκινήσουμε με τις απόψεις μας, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρία λεπτά. Τρία λεπτά, εντάξει, να μας εκθέσει τις απόψεις της. Θα λάβει τον λόγο για τρία λεπτά, παρακαλώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκια και καλημέρα σε όλους. Θα είμαι πράγματι πολύ σύντομη. Λοιπόν, Ουσιαστικά, πέντε από τις έξι χώρες που ανέφερε ο πρόεδρος είναι ασφαλείς, έχουν επικυρώσει, καλύπτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην καταξουσιοδότηση πράξη, οπότε αυτή δεν έχει πια νόημα. Η Κένια ακόμα παραμένει σε κρεμότητα. Ακούσετε τον Υπουργό που έχει κληθεί για το επόμενο σημείο. Προσπαθούμε να έχουμε τις υπογραφές. Ξέρετε ότι υπάρχει σε 8 Σεπτεμβρίου μια διάσκεψη με όλους τους προεδρούς των χωρών ΑΚΕ, οπότε πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και για την περίπτωση της Κένια. Να προσθέσω όμως ότι όσον αφορά τις επικυρώσεις, έχουμε την Αμήβια, την Ποζουάνα, τη Σουαζιλάνδη που έχουν επικυρώσει, αλλά χτες είχαμε πολύ καλά νέα από την Νότια Αφρική. Το Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής ομόφωνα κύρωσε τη συμφωνία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πάντα ε, έμεναν ότι έπρεπε τα κοινοβούλια τους να κυρώσουν και να που γίνεται και αυτό. Επίσης θέλω να πω για τα τεχνικά στοιχεία. Ξέρετε για ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χειριστεί ε, τις ε, προτιμήσεις κτλ. Είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορούμε δηλαδή να μπούμε σε λεπτομέρειες αν θέλετε και διμερώς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητηθεί αυτό εδώ σε όλη την Επιτροπή. Πρόεδρος, υπέροχα, εξαιρετικό, μπράβο και σύντομα. Λοιπόν, από πλευρά εισηγητή για τη Δυτική Αφρική που δεν παρίσταται, ο κύριο Λάμψοφ δεν παρήσατε, αλλά ο κύριο Σόλτ για την Ανατολική Αφρική είναι παρόν, έχει τον λόγο. Κύριε Σόλτ, παρακαλώ. Yep. Μάλιστα. Είχαμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση σε σχέση με την ανταλλαγή απόψεων και όπως όλοι θα γνωρίζετε σε σχέση με την Επιτροπή κάποιες πολιτικές ομάδες έχουν αντιρρήσεις για τέτοιες κατεξουσιοδότηση πράξεις και σε σχέση με την κοινή συζήτηση καθώς εξετάζονται τα θέματα των χωρών της Ανατολικής Αφρικής θα ήθελα να τονίσω αυτή τη συνάντηση, αυτή τη σχέση μια και οι δύο συνάδελφοι δεν μπορούν να εισαγάγουν αυτό το θέμα. Το άρθρο 3 Β και το 23 σε σχέση με την Επιτροπή δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού να αφαιρεθούν κάποιες χώρες από τον κατάλογο των χωρών και σε σχέση με τα όσα έχουν ε, ε, συμβεί. Δεν έγινε όμως αυτό και βρισκόμαστε ας το πω έτσι στην έναρξη σε ε, ισχύ της συμφωνίας και στις 13 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η πρόταση αυτή για έξι κατεξουσιοδότηση πράξης έχει κατατεθεί όπως αναφέρθηκε από εσά Πρόεδρε για έξι ε, χώρες ΑΚΕ αφρικανικές χώρες μεταξύ άλλων. Αυτό, αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνατότητα που μας προσφέρεται να έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στο πλαίσιο των κατεξουσιοδότηση πράξεων που πέρα από τα εμπορικά θέματα έχουν και ευρύτερη εμβέλεια και το θέμα να επιβληθεί μια διορία για τις ε, ε, χώρες ε, για να διασφαλιστεί το τι συμβαίνει ε, πρέπει να δούμε τι, συμβαίνουν, τι σημαίνουν όλα αυτά για μας και για τις χώρες επίσης που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χωρών. Και θα έλεγα ότι εδώ σε σχέση με τα θέματα των κανονισμών αυτών δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, αλλά η ομάδα μας προβληματίζεται πολύ περισσότερο τα πολιτικά ζητήματα και τις πολιτικές επιπτώσεις να λάβουμε υπόψη σε σχέση με τις επιπτώσεις της εφαρμογής τέτοιου είδους κατεξουσιοδότηση πράξεων και για την Κένια και για τα όσα αυτή τη στιγμή διακυβεύονται σε σχέση με την ε, κοινότητα αυτών των χωρών και για κάποιες χώρες της Δυτικής Αφρικής. Μια παρόμοια κατάσταση είχε διαμορφωθεί θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι και πολύ σωστοί και δίκαιοι. Και σε σχέση με την στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις χώρες ε, της ε, Αφρικής, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα δράσουμε και να λάβουμε υπόψη ότι εμείς με τις πολιτικές και εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο να ενδυναμώσουμε τις ε, δικές τους ε, δομές ε, για την περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη ώστε να είναι σε θέση να μπορέσουν περαιτέρω να αναπτυχθούν οι χώρες αυτές. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο με το άρθρο 208 της συνθήκης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την προώθηση όλων των στόχων της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και νομίζω μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε αυτά τα εμπορικά θέματα. Με άλλα λόγια, εμείς η Ενωτική Αριστερά θεωρούμε ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης όπως ε, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τις αρχές της Ένωσης και δεν είναι σωστή μια τέτοια κατεύθυνση και γι' αυτό θα πρέπει κυρίως σε σχέση με τον Οκτώβριο και την προθεσμία μέχρι τον Οκτώβριο να μπορέσουν να αποσυρθούν διότι δεν είναι ρεαλιστικές οι ε, προοπτικές ε, με βάση αυτή την προσέγγιση για αυτές τις χώρες και να δούμε σε σχέση με τις χώρες ΑΚΕ μέσα στην συνάντηση ε, σε σχέση με τον Αϊρόμπι να προσφερθεί μια ευκαιρία να ξαναδούμε τα θέματα των Αφρικανικών χωρών και της Κένιας και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι δεν θα χρειαζόταν αυτή η προθεσμία του ε, διορία του Οκτωβρίου. Πρέπει να δούμε αυτά τα θέματα μέσα σε ένα πλαίσιο ε, δυναμικό, ώστε να μπορέσει ο διάλογος, ο πολιτικός να αναπτυχθεί για την περιφερειακή ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτών των χωρών για την ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε και το τι συνεπάγεται για τις απώλειες όσον αφορά αυτές τις χώρες, ε, ε, ιδιαίτερα και όσον αφορά για παράδειγμα και την Γκάνα. Ευχαριστώ. Για να είμαστε ακριβείς, λέει ο Πρόεδρος, προτείνεται να απορρίψουμε λοιπόν έτσι κάθε μία από αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και να αναβληθεί η προθεσμία για να μπορέσει να διευθετηθεί το θέμα ώστε να έτσι να καλύπτεται αυτός ο στόχος σας. Εντάξει, σωστό, ευχαριστώ. Και τώρα θα λάβουν τον λόγο οι επόμενοι που θέλουν να παρέμβουν από την Επιτροπή μας. Θέλετε να παρέμβετε εσείς, παρακαλώ. Yeah. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή. Ακούσαμε εισαγωγή από το μου θα ήθελα για τη δική μας ομάδα να πω ότι θέλω να επισημάνω ότι οι χώρες για τις οποίες κάνουμε λόγο εδώ όλες δεν είναι λιγότερο ή ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες. Και έτσι για την ομοθεσία που ισχύει υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για διαφορετικές χώρες ε, και ίσως θα ήθελα να ε, πω ότι κάποιοι θα μπορούσαν να θυμούνται εδώ στο Κοινοβούλιο από την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο που είχαμε συζητήσει αυτά. Γνωρίζαμε ότι ε, δεν είναι συμβατά με τον ΠΟΕΠ ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Παρόλα αυτά το κάναμε για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. Υπήρχε ευρύτερη συζήτηση μέχρι πού θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Επί εβδομάδες ανταλλάσσαμε απόψεις μεταξύ των ομάδων και καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό και είπαμε ότι η 1η Οκτωβρίου θα ίσχυε ώστε να έχει χρόνο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουν χρόνο και αυτές οι χώρες για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν. Τώρα το να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο ίσως θα δυσχεράνει το έργο μας στο Κοινοβούλιο και σε σχέση με την προθεσμία του Οκτωβρίου αν μετατεθεί για 1,5-2 χρόνια αργότερα αυτή η ημερομηνία. Γι' αυτό θα ήμουν ευγνώμων αν κάναμε κάθε προσπάθεια τις χώρες αυτές που αφορώνται εδώ και καλούνται ε, σε σχέση με αυτά να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους ναι, για τις συμφωνίες αυτές που ε, καθώς θα έχουν υπογραφεί θα διασφαλίζουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα πρέπει όμως να στείλουμε λάθος μηνύματα με μεταβάλλοντας και αναβάλλοντας την προθεσμία. Συμφωνήσαμε 1η Οκτωβρίου 2016. Αν δούμε ποιες χώρες εδώ θα πρέπει να υπογράψουν και τα προβλήματα που υπάρχουν πρέπει να δούμε και να αναγνωρίσουμε ότι τα προβλήματα γι' αυτό θα πρόκειται για μια ή δύο χώρες στο τέλος τέλος που ουσιαστικά δεν μπορούν να ε, θέσουν όσο ομήρους στις υπόλοιπες χώρες και σε σχέση με τη μετάθεση της προθεσμίας θα δημιουργούν το πρόβλημα. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η δική μου η ομάδα έχει αντίρρηση για αυτές τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση. Ε, η Σάντρα ήταν ιδιαίτερα ε, λακωνική, αλλά θα ήθελα να μας πει λίγο περισσότερα και να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις, κυρίως για την Μποτσουάνα και τη Ζουαζιλάνδη. Ε, δεδομένου των όσων ακούσαμε, διότι το υπονόησε, αλλά δεν μας το είπε ακριβώς, ε, αν σκοπεύετε ε, να αποσύρετε την πράξη κατά εξουσιοδότηση για αυτές τις χώρες. Θα αποσυρθεί η πράξη εξουσιοδότηση, οι συγκεκριμένες δηλαδή αναχώρα. Όσον αφορά την ECOWAS, αυτό ακόμα ε, δεν το έχουν υπογράψει όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Η Γκάνα δεν έχει υπογράψει την ε, ενδιάμεση ε, σύμβαση του 2007 αυτό σημαίνει ότι θα αποσυρθεί αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση ή αν υπογραφεί η ε, συμφωνία του 2014 ε, θα υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης, διότι νομίζω ότι αυτό θα ήταν άδικο για την ακτή του Ελεφαντιστούν και την Κάνα ε, να τιμωρούνται παρά το γεγονός επειδή μάλλον δεν έχουν υπογράψει σε διάμεσες συμφωνίες. Ο κύριος Σόλτς έχει απόλυτα δίκιο η Κένια είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Η Κένια βέβαια έχει κάνει ό,τι μπορεί, έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να υπογράψει τη Συμφωνία ε, Ελευθέρων Συναλλαγών, αλλά ουσιαστικά την έχουν απογοητεύσει οι εταίροι της. Και γιατί σε αυτή την περίπτωση να πρέπει να τιμωρείται η Κένια. Εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιπόν μια πράξη κατεξουσιοδότηση για την Κένια δεδομένων των συνθήκων. Για να μη μακρηγορώ να πω ότι ο Χέλμουντ Σόλτς ε, ε, είχε ένα πολύ σωστό επιχείρημα. Ε, νομίζω ότι η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου δεν είναι ρεαλιστική. Υπάρχει κάποιο επιχείρημα για να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και να έχουμε μια πιο λογική προθεσμία για αυτές τις χώρες. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, διότι χρειαζόμαστε ένα σοβαρό στόχο και η 1η Οκτωβρίου δεν είναι σοβαρό στόχος. Μετά από την ε, παρέμβαση των άλλων μελών θα σου δώσουμε λόγο για να απαντήσεις. Ε, η Σκακέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πολύ για τη μικρή καθυστέρηση. Αλλά έχω μια εικόνα του τι είπατε. Νομίζω ότι και για μας θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις, όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι. θα αποσύρετε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ποιες ε, και ποιος έχει υπογράψει τι, ποιος έχει υπογράψει ενδιάμεσες συμφωνίες ε, και ποιος έχει υπογράψει ε, την τελική συμφωνία. Και επίσης κυρίως όσον αφορά την ECOWAS, εμείς έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα εν γέννη. Το όλο θέμα θα πρέπει να είναι να λάβουμε υπόψη μας και ποια είναι η πιο λογική οικονομική δομή ε, για τις χώρες αυτές. Δεν είναι βέβαια μόνο δική μας δουλειά αυτή, είναι και δική τους δουλειά, αλλά η περιφερειακή οικονομία είναι από τα θέματα τα οποία συνεχώς επισημαίνονται. Και αν κάποιες χώρες συμμετέχουν στην ΕΚΟΓΟΣ και κάποιες άλλες δεν συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν αργότερα, αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΚΟΓΟΣ. Το αυτό ισχύει και για άλλες ε, συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλακών. Στην αρχή ήταν υποτίθεται περιφερειακή συμφωνία, μετά έμενε μια χώρα έξω και αυτό φυσικά έχετε να ζημιώσει την περιφερειακή οικονομία και εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε πλήρη συμμετοχή και να το εξετάσουμε και από το πρίσμα της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη, η οποία λογικά θα έπρεπε να προωθείται. Συμφωνώ επίσης με τους ε, συναδέλφους όσον αφορά το θέμα της προθεσμίας. Η ομάδα μου ποτέ δεν πίστευε ότι μπορεί να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Ε, συνήθως όταν θέτουμε προθεσμίες δεν λειτουργεί το σύστημα, είναι πιο περίπλοκα. Για την περίπτωση της Κένιας ακούσαμε ήδη τι συμβαίνει. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε πιο ρεαλιστικές προθεσμίες και να μην ε, το χρησιμοποιούμε ως ε, εκβιασμό δεν είναι ε, πολιτικό εργαλείο εκβιασμός, αλλά τελικά τίνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Και θα πρέπει να θυμάστε ότι το θέμα της 1ης Οκτωβρίου ήταν ένα πολιτικό θέμα, το οποίο δεν βασίστηκε σε ρεαλιστικές προσδοκίες, αλλά περισσότερο σε πολιτική κληρονομιά. Ευχαριστώ, η Έμα. Να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως ε, την ε, διαδικασία και θέλουμε όλες οι χώρες ΑΚΕ να έχουν ε, στεναρή, ισχυρή νομική βάση. Ε, και είναι κρίμα που ακούμε ότι κάποιες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής έχουν ε, δυσκολίες μετά από τη σύναψη των συμφωνιών, κυρίως όσον αφορά την Κένια η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θα χάσει τις προτιμησιακές δυνατότητες που έχει για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, ε, καλό ήταν να έχουμε αυτές τις πράξεις εξουσιοδότηση. Ε, θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται αν η κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής δεν υπογράψει τη συμφωνία και τι γίνεται με την ε, συμφωνία της ε, Δυτικής Αφρικής εάν οι χώρες αρνηθούν να υπογράψουν. Ε, και θα θέλαμε περισσότερα και από τις χώρες αυτές. Είναι συμφωνία εταιρική σύμπραξη αυτή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές. Αν υπάρχει λοιπόν μια ευκαιρία ε, να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεω. καλό θα ήταν να γίνει. Μαρία Ρένα, ευχαριστώ. Θλίβομαι για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματικά και λυπάμαι γιατί έρχεται πολύ κακή στιγμή μετά από πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις τρεις διαφορετικές αφρικανικές περιφέρειες και έχουμε την αίσθηση ότι η τακτική αυτή της Επιτροπής είναι προκειμένου να υποχρεώσει ορισμένες χώρες να θέσουν υπό αμφισβήτηση συζητήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των συζητήσεων. Πρέπει να δουλεύουμε στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι αστάθεια στις οικονομίες εκείνες οι οποίε έχουν τάση να ενισχύονται στην Αφρική, Κένια για παράδειγμα, και ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Κένιας που είναι εδώ σήμερα. Είναι μια οικονομία η οποία διαφοροποιείται σήμερα και με το χτύπημα αυτό ε, στην Κένια, ενώ προσπαθεί. Γιατί θυμόσαστε ότι στην αρχή δεν ήταν υπέρ των συμφωνιών αυτών, ενώ τώρα είναι. Οπότε δημιουργείται μια ομοιρία, παίρνουμε όμοιρο την Κένια με αρνητικά αποτελέσματα. Η στάση αυτή της Ευρώπης για μένα είναι απαράδεκτη. Επίσης, κάποιες χώρες και κυρίως η σχέση Ευρώπης-Αφρικής οδηγείται σε έλλειψη εμπιστοσύνη. και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα με την Αφρική δεν έχουμε μόνο οικονομικές σχέσεις. Όλες οι σημερινές συζητήσεις για τη μετανάστευση που μας έρχεται από την Αφρική έχει να κάνει και με τον οικονομικό παράγοντα. Τι κάνουμε δηλαδή οικονομικά. Ζητάω λοιπόν περισσότερη συνοχή ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Αφρική και όχι μόνο μια πολιτική περιορισμών απέναντι στις αφρικανικές χώρες. Έπειτα μιλάμε πάντα για λογική προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Τι είναι αυτό όμως το Ντελέρε Έχουμε μιλήσει για περιφερειακές συμφωνίες και μετά όταν είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για τις περιφερειακές αυτές συμφωνίες, κάναμε προσωρινές διμερείς συμφωνίες με την Κάνα, για παράδειγμα. Και στις περιφερειακές συμφωνίες ξαναβάζουμε αυτό το λογικό χρονικό διάστημα. Μα μιλάμε για τις περιφερειακές συμφωνίες Νότου, Ανατολής κτλ. ή για τις διμερείς συμφωνίες. Θέλω να μου το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εγώ βλέπω κάποιο χάος. Μας λένε ότι υπάρχει προσωρινή συμφωνία με την Γκάνα. Ναι, η Γκάνα δεν εξαιρείται. Οπότε εγώ δεν έχω καταλάβει για τι πράγμα μιλάνε. Δεύτερον, όταν μιλάμε για αυτήν τη λογική προθεσμία, είναι αλήθεια ότι για την Νότια Αφρική τηρούμε τις προθεσμίες, δηλαδή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 13 Σεπτεμβρίου, στην Ολομέλεια δηλαδή, μπορούμε τότε να τηρήσουμε την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου για πρόσβαση στις αγορές των χωρών εκείνων που περιλαμβάνονται στις κατεξουδότηση πράξεις όπως είναι η Ναμίδια. Όμως όσον αφορά την Ανατολή και τη Δύση, δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία για ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι τιμωρούμε τις αφρικανικές χώρες ουσιαστικά επειδή εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε προθεσμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνει, προβλέπει οι συμφωνίε αυτέ οι περιφερειακέ να ψηφιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης κύριε Κασπαρή να γνωρίζετε ότι πριν από δύο χρόνια ναι, υπήρξε μια συμφωνία, αλλά στο μεταξύ άλλαξαν πολλά. Και νομίζω ότι η πολιτική κατάσταση στον Μπουρούντι σχετικά με την συμφωνία με την Ανατολική Αφρική θέτει πρόβλημα για τους Ευρωπαίους προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία με μια χώρα η οποία παραβιάζει πλήρως τις συμφωνίες του Κατονού. Η κυρία Ντερινή έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού και Άρα δεν είναι δυνατόν εμείς Ευρωπαίοι να ψηφίσουμε μία συμφωνία για την οποία το άρθρο 96 έχει ενεργοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να υπάρχει συνοχή. Πριν από δύο χρόνια η κατάσταση στον Μπουρούντι ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άρθρο 96 έχει ενεργοποιηθεί και άρα δεν μπορούμε να υπογράψουμε, να υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να μπει τάξη στην πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Trade όσον αφορά την Αφρική. Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου. Επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ βρίσκω ότι η κατεξουσιοδότηση νομικές πράξεις είναι ένα τυχέστατο μέσο. Αντιφάσκει στο πνεύμα μιας εταιρικής σχέσης σε μια εταιρική σχέση προσπαθεί κανείς από κοινού να προχωρήσει παραπέρα και χωρίς ε, κάποια τέτοια πίεση. Και είναι μια μηχανιστική νοοτροπία που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Τώρα, να μπορεί κανείς να πει τώρα τέρμα πια τελεία και παύλα είναι κατανοητό αυτό για κάποιες περιπτώσεις και να πούμε ότι για μια, για μια περίοδο δύο ετών αποφασίστηκε μια τυπική διαδικασία που θα πρέπει να ισχύει. Έχει δίκιο η κυρία Ρένα ότι κάποια πράγματα πρέπει να ε, ισχύουν κάποια πράγματα. Όμως σε πολλές προθεσμίες δεν τηρήθηκαν. Γι' αυτό είμαστε κατά των κατεξουσιοδών της υπράξεων που αντιφάσκουν. Δεύτερον, είναι απόλυτα περιτές. Περιτές και στις χώρες εκείνες όπου υπάρχουν προβλήματα είναι προβλήματα που με κατεξουσιοδότηση πράξη ε, δεν μπορούν να επιληθούν. Και πρέπει πολιτικά να προβληματιστούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βοηθηθούν οι χώρες αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν ή να απορριφθούν αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις ή να αφαιθεί ανοιχτή η διαδικασία να απορριθουν αυτες οι κατεξουσιοδοτηση πραξεις η να αποσυρθούν. Γιατί σε ένα κλίμα εταιρική σχέση δεν μπορούμε να ασκούμε πιέσει ε, και να απειλούμε με τέτοιου είδου κατεξουσιοδότηση πράξη και να επιδεινώνουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Έχετε τώρα την ευκαιρία να απαντήσετε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για όλες τις ενδιαφέρουσες αυτές ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι περίπλοκο το θέμα, οπότε θα προσπαθήσω να ξεμπερδέψω κάπως τα τεχνικά στοιχεία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε διευκρινίζοντας ότι ο τελικός μας στόχος είναι το περιφερειακό. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Κάποιες ε, είναι λιγότερο τέλειες λύσεις. Η Γάνα, το αλεφαντοστού πρέπει να κρατήσουν το προτιμησιακό καθεστώς τους και το επέλεξαν με αυτό που ονομάζουμε Stepping Stone Agreement. Τώρα για μας η περιφέρεια είναι ο στόχος. Δεν παρετούμεθα από αυτόν. Αλλά έχω καταλάβει ότι οι συμφωνίες αυτές εταιρικές σχέσης είναι κάτι σταδιακό δεν φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα έτσι με μιας. Λοιπόν, ξεκινάμε από την επικύρωση μιας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Έχετε μια ε, τέτοια συμφωνία, την κυρώνετε και μετά προχωρούν τα πράγματα. Τώρα, αυτοί που είναι τυχεροί και έχουν μια προσωρινή τέτοια οικονομική εταιρική σχέση, όπως η Γκάνα, θα μπουν στο καθεστώς αυτό ΣΟΕΣ. Από την αρχή. Από την άλλη όμως, αυτές που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως η Κένια, κυρώνοντας αυτή την περιφερειακή συμφωνία, Έτσι καλώς αν έχουμε τις πέντε υπογραφές και τις πέντε κυρώσεις, η οικονομική εταιρική ε, σχέση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από την οικονομική εταιρική σχέση και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Τότε το προτιμησιακό καθεστώς συνεχίζεται. Πρέπει όμως επίσης να πω ότι οι προθεσμίες μπορεί να αιτιολογούνται πάντα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και ολόκληρη την εικόνα. Αυτό που κάνουμε δίνοντας ε, πλήρη ελεύθερη πρόσβαση σε ποσοστώσεις σε αναδυόμενες οικονομίες που είναι δυνατές, ε, αυτό το βλέπουν και οι άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ και κάνουν τις συγκρίσεις τους. Η Βολιβία δεν έχει τα ίδια επίπεδα με τις αφρικανικές χώρες τις οποίες αναφερόμαστε τώρα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν τους δώσουμε πλήρη απελευθέρωση ποσοστώσεων, ενώ υπάρχουν άλλες που δεν έχουν το ίδιο καθεστώς, αν το κάνουμε αυτό πρέπει στα πλαίσια του ΠΟΕ να υπάρχει κάποια συμβατότητα. Για τις έξι αυτές θα έλεγα ότι πέντε από τις έξι έχουν τέτοια βάση στον ΠΟΕ. Η Κένια όμως παραμένει εκτός μετά την κύρωση αυτών των ε, εταιρικών ε, σχέσεων του 2014. Εμείς δίνουμε την επιλογή στις χώρες, γιατί είναι αυτό ή το GSP. Το GSP είναι επίσης μια επιλογή γενικευμένες ε, προτιμήσεις. Όμως επιμένουμε ότι τα κοινοβούλια έχουν αποφανθεί. Τα κοινοβούλια των χωρών έχουν αποφασίσει τι δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν και τι οικονομικό καθεστώς θέλουν να ακολουθήσουν. Άκουσα την άποψη της κυρίας Κέλλερ. Είναι επιλογή τους. Πιστέψτε το, μετά από 12 χρόνια δεν υπάρχει μεγάλη πίεση. Η προθεσμία που έχει επιλέξει την 1η Οκτωβρίου δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν επενθυμίσω το Κοινοβούλιο ήθελε 1η ε, Οκτωβρίου 2016. Δεν θέλω να το κάνω θέμα πάντως. Κατά σύμπτωση εδώ έχουμε φτάσει. Λοιπόν, για πέντε χώρες δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχουν επιλέξει. Περιφερειακά εξακολουθούμε να θέλουμε να έχουμε περιφερειακή συμφωνία. Και καμία χώρα δεν είπε ότι δεν θα υπογράψει ΣΟΕΣ. Η Νιγηρία θέλει να προχωρήσει, αλλά έχει πολλά ζητήματα ακόμα. Η κάθε χώρα, λοιπόν, λοιπόν έχει το δικό της ρυθμό για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Να είμαστε όμως ξεκάθαροι ότι η επιλογή χωρών όπως Ελεφαντοστού και Γκάνα συνάδουν με το γεγονός ότι θέλουν να έχουν ισχυρές σχέσεις με τον μεγάλο εταίρο και από πλευράς εμπορίου και από πλευράς ανάπτυξης. Δεν βλέπουν μέλλον χωρίς την Ευρώπη. Καλό είναι αυτό για μας. Τους ενδιαφέρουμε. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό να ισχύει όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για άλλους τομείς. Ανθρώπινα δικαιώματα, εφόρος ανάπτυξη κλπ. κλπ. Είπατε ότι τιμωρούμε κάποιες χώρες. Όχι. Όντως μερικές φορές η λύση δεν είναι η τέλεια, αλλά ο τελικός στόχος είναι η περιφερειακή συμφωνία. Και σε αυτές τις χώρες προσφέρουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν μια καλή σχέση μαζί μας. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι άλλοι δεν έχουν αυτήν την προνομιακή σχέση, παρόλο που μπορεί οικονομικά να βρίσκονται, ε, να έχουν πολλά κοινά. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας, αλλά εδώ είμαι, στη διάθεσή σας. Πρόεδρος. Με τις κατεξοδότηση πράξη θα κάνετε, θα τις αποσύρετε. Δεδομένου ότι δεν έχουν πια νόημα, θα τις ε, αποσύρουμε προφανώς. Να σας πω και τις ημερομηνίες κύρωσης Μποτσουάνα 30 Ιουνίου. Τα μέσα που έχουν ε, υποβληθεί έτσι. Ακτή Ελεφαντοστού 12 Αυγούστου, Γκάν 3 Αυγούστου, Κένια δυστυχώς όχι ακόμα, Ναμίβια 6 Ιουλίου και Σουαζιλάνδη 26 Αυγούστου. Και περιμένουμε την κύρωση της Νότιας Αφρικής που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Ο Χέλμουτ. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και έχω επιπρόσθετη ερώτηση προς εμάς. Επειδή κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την Κάνα και την ακτή ελεφάντος του αναφέρονται στην εταιρική συμφωνία του 2014. Δηλαδή θα πάνε σε μια προσωρινή ενδιάμεση τώρα συμφωνία ε, ε, ε εταιρικής οικονομικής σχέσης. Περί τίνος γίνεται λόγος ε, τώρα εδώ γιατί διαφορετικά δεν θα ε, γνωρίζουμε, δεν θα ε, ε, μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Ποια είναι τα θέματα λοιπόν της κατεξουσιοδότησης πράξης εδώ να επαναλάβω ότι ε, το έναυσμα είναι η κύρωση μιας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Θα δείτε ότι στην πράξη κατά εξουσιοδότηση, να τη διαβάσετε προσεκτικά, δεν γράφουμε ποτέ ότι πρέπει οπωσδήποτε να κυρώσετε αυτή τη συμφωνία, γιατί τότε θα ήταν μια πράξη κατά που είναι περιττή, γιατί αυτό ισχύει στην πραγματικότητα, η κύρωση της περιφερειακής συμφωνίας. Αυτή ε, θα αποτελέσει ε, γεγονός για τη Δυτική Αφρική, ε, είναι αυτό το οποίο ε, ξεκινά τη συμφωνία του 2014. Τώρα, το κατά πόσον ε, μία χώρα μεμονωμένα διατηρεί το προτιμησιακό της καθεστώς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αντικείμενο της πράξης κατά εξουσιοδότηση. Νομίζω ότι ε, δεν συζητάμε απαραίτητο να υποχρεώσουμε κάποιες χώρες να παραμείνουν σε ένα μέσο που δεν επιθυμούν. Εάν όμως επιθυμούν να παραμείνουν ε, στο προτιμησιακό καθεστώς και δεν θέλετε ε, το GSP, είστε διατεθειμένοι να συμμετέχετε σε αυτή τη συμφωνία. Και επιμένω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε μια ε, εύρωστη νομική βάση ενώπιον του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ δεν έχει καμία αντίρρηση για τη συμφωνία με την Κάνα, αλλά εάν δεχτούμε την Κένια θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, θα πρέπει δηλαδή να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι θέμα προθεσμιών. Συμφωνώ, οι προθεσμίες είναι επώδυνες, αλλά είναι θέμα δικαιοσύνης. Ε, θα γίνει και ένα πρόγευμα για το ε, θεμητό και δίκαιο εμπόριο. Ε, πρέπει να υπάρχει λοιπόν και ισότιμη μεταχείριση για κάθε χώρα. Και επαναλαμβάνω ότι για μα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε ενώπιον αυτών των χωρών και πέραν ε, του εμπορίου. Ε, αυτό βέβαια δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ε, πολλοί αναφέρθηκαν στη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Αφρική και τη σχέση μεταξύ των και λογικά είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία έχουμε με αυτές τις χώρες που πρέπει να υπάρχει κάτι πέραν του εμπορίου. Αλλά κάνω έκκληση, δεχτείτε ε, ε, την επιλογή αυτών των χωρών να υπάρχει αυτή η προσωρινή λύση που δεν είναι και η βέλτιστη δυνατή ε, και όπως είπα εγώ είμαι ακόμα αισιόδοξη για τη συμφωνία. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν να υπογράψουν. Μια επιπλέον ερώτηση από την κυρία Κερτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου, Σάντρα. Θέλω όμως να είναι απόλυτα σαφές και σας παρακαλώ απαντήστε με ένα ναι ή όχι είπατε ότι οι πέντε καταξουσιοδότηση πράξεις πλέον ε, είναι περιτές. Και επειδή έχουν υποβληθεί επισίδων, όμως δεν πρέπει να γίνει μια επίσημη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόσυρση αυτών των πράξεων καταξουσιοδότηση. Θα τις αποσύρετε, ναι ή όχι. Ναι. Και το είπα και για να σας προλάβω. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι απαιτείται. Ωραία, θα ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση για τις πράξεις κατεξουσιοδότησης εδώ, στην Επιτροπή. Θα αποφασίσουμε επί της διαδικασίας ε, στην ε, ε, συνάντηση των συντονιστών αργότερα. για τη Συμφωνία για την Ανατολική Αφρική. Θα συνεχίσουμε με το σημείο που έχουμε στη συνέχεια, στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω το λόγο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 στις ίδιες ομάδες εργασίας ε, στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΟΕ. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο και προς όλα τα μέλη της Επιτροπής σας, διότι μας δώσατε αυτή τη δυνατότητα και όπως γνωρίζετε, στην Ασία αυτή τη στιγμή ξεκινάει η οικονομική ασιατική κοινότητα η οποία ε, βλέπει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ακριβώ είμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Θα θέλαμε η Ινδονησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια διμερή ομάδα φιλίας. Όπως γνωρίζετε, η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα στην ΑΣΕΑΝ και η έδρα της ΑΣΕΑΝ είναι στη Τζακάρτα, στην Ινδονησία. Επομένως, πραγματικά ε, ελπίζουμε να υπάρχει μια ομάδα φίλων Ινδονησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις ε, ε, σχέσεις Ινδονησίας ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Θα συναντηθούμε και με τους εταίρους μας ε, από το Βελγικό Κοινοβούλιο και θα δούμε και το, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αρμόδια για θέματα εμπορίου. Ε, είμαστε μια ε, πολυάριθμη αντιπροσωπεία και έχουμε έρθει από χθε. Να σας ευχαριστώ. Είναι εδώ και ο πρέσβης μας, ο Ινδονήσιος, ο Ινδονήσιος πρέσβης εδώ και φυσικά και το προσωπικό μας. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φιλία μας και φυσικά το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ Ινδονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η Έμα θέλει να κάνει ένα σύντομο... Η Μακουλάδα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να καλωσορίσω την αντιπροσωπή από την Ινδονησία εδώ. Οι δεσμοί είναι πολλοί μεταξύ μας. Στον ΠΟΕ, μεταξύ άλλων, και πρέπει να τους ενισχύσουμε προκειμένου η συμφωνία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας να είναι μια συμφωνία, να καταλήξει μια συμφωνία καλή, όπου οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας να βοηθήσουν να ενισχυθούν οι σχέσεις μας και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών μας αλλά και η ζωή των εργαζομένων μας. Ευχαριστώ λοιπόν και θέλω να πω στην επικεφαλής αντιπροσωπείας που είναι και γυναίκα. Θα δουλέψουμε και για τον ρόλο των γυναικών για να βελτιωθούν οι ευκαιρίες που έχει το 50% του πληθυσμού. Και συμφωνώ και εγώ για τη δημιουργία αυτής της ομάδας φιλίας μεταξύ Ευρωβουλευτών και Βουλευτών της Ινδονησίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία και προσβλέπουμε καλή συνεργασία στο μέλλον μεταξύ μας. Εντάξει συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 11. Ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ανατολική Αφρική. Αρκετές φορές το έχουμε αναφέρει. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά ακριβώ για αυτό, με τα διάφορα προβλήματα τα οποία συνδέονται με αυτό το ζήτημα. στις 16 Οκτωβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η υπογραφή προβλεπόταν για τον Ιούλιο 2016 στο Ναϊρόμπι στην Σύνοδο εκεί όμως αναβλήθηκε αναβλήθηκε επειδή η Τανζανία δεν υπέγραψε ή δεν ήθελε να υπογράψει και τελικά έχουμε τώρα το πρόβλημα ιδιαίτερα για την Κένια ως μόνο μη ανεπτυγμένο κράτος σε σχέση με άλλα ότι χωρίς αυτή την ε, εμπορική εταιρική συμφωνία θα μπορούσε να απολέσει την πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε τώρα εδώ ως θέμα. Χαίρομαι για το ότι και ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου της Κένια παρίσταται, είναι εδώ παρόν στην αίθουσα. Καταρχήν ο εισηγητής Σόλτς θα λάβει τον λόγο και μετά ο κύριος Υπουργός Εμπορίου από την Κένια. Παρακαλώ κύριε Σόλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και καλωσορίζω και εγώ θερμά τον Υπουργό Εμπορίου της Κένιας ανάμεσά μας. Παρακολουθώντας αυτό το πολύ θα έλεγα υψηλών προκλήσεων θέμα θα ήθελα να τονίσω εισάγοντας αυτό το θέμα με μια μικρή αναδρομή. Εδώ μπορεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία όταν οι πέντε εμπλεκόμενες χώρες Ουγγάντα, Κένια, Τανζανία που ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες η Ρουάντα και το Μπουρούντι προστέθηκαν στη συνέχεια και το Νοέμβριο 2007 υπήρξε το πλαίσιο λοιπόν για αυτές τις διαδικασίες ε, που εγκρίθηκε. Οι χώρες αυτές θα ήθελαν πλήρως να διαπραγματευτούν την περιφερειακή αυτή εμπορική εταιρική σχέση και προχώρησαν σε σχέση με την Προεδρική Επιτροπή ε, λαμβάνοντας υπόψη κάποια επίμαχα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν ιδιαίτερα θέματα τα οποία αφορούν ε, ζητήματα πολιτικής ε, και ζητήματα ε, εμπορικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε και ένα ψήφισμα του 2009 για αυτή την προσωρινή συμφωνία. Θα ήθελα να αναφέρω τρία παραθέματα από αυτό το ψήφισμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει επαρκή και ε, ε, διευρυμένη σύνδρομη σε αυτές τις χώρες ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των οικονομιών τους μετά την υπογραφή αυτής της ε, εμπορικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προτείνεται να υπάρξει προσέγγιση και επικέντρωση σε σχέση με τα γεωργικά αγαθά ώστε να μπορέσουν να προστατευθούν οι βιομηχανίες, οι ε, οικονομίες αυτών των χωρών όπως θα έπρεπε. Και ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ο κέριος ρόλος ε, της ε, Συνόδου των Κοινοβουλίων και ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίζει την εμπλοκή αυτών των χωρών και αυτών των θεσμικών οργάνων στο μέλλον και καλή σε σχέση με τις χώρες αυτές να υπάρξει αυτή η προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε την προσέγγιση αυτή όπως έχουμε καταλήξει σήμερα, όπως έχουν καταλήξει τα πράγματα, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η εμπορική εταιρική συμφωνία. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει επιτευχθεί μια πραγματική έντονη, ενδυναμωμένη ολοκλήρωση περιφερειακή ώστε να υπάρξει μια παγιωμένη, ένας ε, ε, αποτελεσματικός τρόπος και διαδικασίες συνεργασίας ήδη ξεκινώντας το 2005 με μια πλήρη ανάπτυξη ε, στη συνέχεια αυτών των δυνατοτήτων. Και τον Νοέμβριο 2013 για παράδειγμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο που ε, ε, θα υπεγράφεται. έγιναν όλες οι διαδικασίες, όλα τα διαβήματα ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι χώρες αυτές μέσω της περιφερειακής αυτής εμπορικής εταιρικής σχέσης να προσχωρήσουν προς αυτές τις δυνατότητες. Και επίσης σε σχέση με το να ζητηθεί για παράδειγμα ε, όταν από το ε, ε, Σουδάν ζητήθηκε με το αντίστοιχο άρθρο της ΙΠΑ να δημιουργηθεί η δυνατότητα να μπορέσουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης να ενταχθούν σε αυτή την εταιρική σχέση. Είναι μια υποεξέλιξη λοιπόν διαδικασία. Αναφέρθηκε ήδη το θέμα ότι αποτελείται από, έχουμε τον Μπουρούντι, τη Ρουάντα, την Τανζανία, την Ουγκάντα, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και την Κένια, που ε, σε σχέση με το καθεστώς τους ως ε, μελών του ΠΟΕ, η μη επικύρωση της συμφωνίας μέχρι τον Οκτώβριο θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, για τις χώρες αυτές, ιδιαίτερα όμως για την Κένια. Και νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στο, από πλευρά σας συντονιστών πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το τι σημαίνει αυτό να μην έχουν ε, τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις σε πέντε χώρες και να απομένει μια χώρα ε, σε εκκρεμότητα χωρίς να έχει ρυθμίσει αυτά τα θέματα και προβλήματα σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά ε, που δημιουργούνται για τις άλλες χώρες αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα και μπορεί να υπάρχει μια χωρίς ποσοστώσεις δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές ε, εφόσον συμμορφώνονται. Περνάω τώρα στα σχέση με τις πτυχές των εμπορικών σχέσεων, εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα αυξανόμενο πλαίσιο και ε, όγκων ε, βλέπουμε και το ποσοστό ανάπτυξη ήταν 14,4% για τις εισαγωγές σε σχέση με τις ε, ε, χώρες αυτές 5% και το 2015 οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ και τα εισαγόμενα ήταν 2,6 αξίας 2,6 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό σημαίνει για το συνολικό εμπόριο έχουμε μία διαφορά σε σχέση με τις εισαγωγές-εξαγωγές. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να μην θεωρηθεί, δεν είναι ένα σημαντικό μέγεθος αυτό, έχει όμως επιπτώσεις για τις χώρες αυτές και για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανάγονται σε ένα υψηλό ποσοστό, για παράδειγμα έχουμε και το 3% ε, για παράδειγμα εισαγωγών των προϊόντων συνολικά. Αν δει τις λεπτομέρειες και δει κανείς και το δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κατανοήσουμε όλες τις επιπτώσεις ε, ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών σε περίπτωση αποχώρησής του λοιπόν για τις ε, εμπορικές σχέσεις ε, και τη διαμόρφωσή τους σε σχέση με τις χώρες της Αφρικής. για τις πιο σημαντικές εξαγωγές της Κένιας για παράδειγμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό 57,8% του συνολικού 178 δισεκατομμυρίων ένα γεγονός το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη το συμπέρασμα, το, η σύναψη της ε, εμπορικής εταιρικής σχέσης και σε σχέση με τις ε, εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις από τον Οκτώβριο του 2014 που δόθηκε η παράταση από εκείνη την ε, ημερομηνία ε, ε, οι εξαγωγές για παράδειγμα της Κένιας ιδιαίτερα των <clears throat> λουλουδιών από την Κένια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σημαντικότατες επιπτώσεις ε, για τον παραγωγικό τομέα ε, και την ε, οικονομία της Κένιας λόγω αυτής της κατάστασης. Η κατάσταση το 2015 οδήγησε το Συμβούλιο στο να μπορέσει μέσω της υπογραφής της προσπάθειας ε, να ρυθμιστεί το θέμα με μια συμφωνία που θα υπογραφόταν τον ε, Ιούλιο εκκρεμεί ακόμα και επίσης θέλω να αναφέρω για άλλη μια φορά το πρόβλημα του Μπουρούντι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το περίπλοκο θέμα για το που έχουμε καταλήξει σε σχέση με όλα αυτά και να δούμε τι σημαίνει υπό την πολιτική ετοιμότητα και προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να προχωρήσει στο να λάβει υπόψη και να ε, σταθμίσει ε, τις πολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ε, στάσης από πλευράς της θα έχουμε και την έκθεση που θα ε, παρουσιαστεί, ε, θα κατατεθεί αναμένοντας φυσικά την ε, περαιτέρω εξέλιξη αυτού, αυτού του θέματος. Επί της ουσίας, από πλευράς περιφέρειας προς περιφέρεια και το τονίζω αυτό, είναι μια συμφωνία που καλύπτει περιφέρειες σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις και την οικονομική συνεργασία. Τονίζεται η σημασία, η σπουδαιότητα της απελευθέρωσης των διαδικασιών πρόσφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απελευθέρωση από ποσοστώσεις και αναλήφθηκε η υποχρέωση να υπάρξει απελευθέρωση για μια 25 ετή περίοδο των ε, διαδικασιών για συγκεκριμένα προϊόντα και σε σχέση με ε, για παράδειγμα ε, χημικά προϊόντα ή κλωστοϊφαντουργικά να υπάρξει μια σχετική διαμόρφωση προσαρμοσμένη στις ανάγκες πράγμα το οποίο θα λάμβανε υπόψη τις ανάγκες και σε περίπτωση διατήρησης των περιφερειακών προτιμήσεων θα έπρεπε περαιτέρω να υπάρξει δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η ε, εμπορική εταιρική συμφωνία ώστε να υπάρξει η αναγκαία ελαστικότητα, η αναγκαία ευληγησία ώστε να υπάρξουν και οι αναγκαίες ρήτρες διασφάλισης ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εισαγωγών πράγμα το οποίο θα δίνει την δυνατότητα με τον ε, πιο εύθετο τρόπο να προστατεύονται αυτά τα αγαθά. Σε σχέση με την μη εφαρμογή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτήσεων ή ενισχύσεων όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα ή την εξαγωγή τέτοιων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που υπάρχουν υπάρχει και ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά την συνεργασία για την ανάπτυξη και την ταυτοποίηση των οικονομικών αναγκών και την ρύθμιση σε σχέση με τους εταίρους. <clears throat> Από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην μακρηγορήσω θέλω να υπογραμμίσω ένα σημαντικό θέμα που ανήκει και αυτό μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης, ε, στο πλαίσιο της ακρόασης. Σε σχέση με τη Συμφωνία Κοτονού για την αηφορία της ανάπτυξης ε, που δεν υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σχετικά που θα λέγα ότι θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί εδώ πρέπει να μπορέσει να συμπεριληφθεί υπό την μορφή ρητρών και μια ρήτρα που θα αναφέρει, αναφέρεται στη Συμφωνία Κορτονού είναι ε, σημαντικό θέμα όπως και η αναφορά και η λήψη υπόψη του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των αντίστοιχων διαδικασιών. Και Φυσικά σε σχέση και με την ακρόαση αυτή θέλω να πω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τις συζητήσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη σε σχέση με τις χώρες αυτές για τον στόχο και την κατεύθυνση αυτής της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις χώρες αυτές. Και έχουμε και παρόμοιες αντίστοιχες συζητήσεις εμείς εδώ για την κατεύθυνση και το εύρος αυτών των θεμάτων θα υπάρχει αναθεώρηση, επανεξέταση σε πενταετής περιόδους και μέσω των κοινών θεσμικών οργάνων όπως και του Συμβουλίου της, για τα θέματα εταιρικών εμπορικών σχέσεων και ε, ε, επίσης σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δούμε πώς τα σώματα, οι φορείς που θα εποπτεύουν την εφαρμογή και υλοποίηση όλων αυτών θα μπορούν να ε, δρούν ώστε να ε, προσαρμόζονται στις ε, ανάγκες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα στη συνέχεια. Το στοιχείο το οποίο αφορά το χρονοδιάγραμμα και το οποίο έχει καθοριστεί και θα αφορά και τις ανταλλαγές απόψεων πρέπει να αναμείνουμε ώστε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από πλευράς μας. Πρέπει να αναμείνουμε τις περαιτέρω εξελίξεις που βρίσκονται εν ρευστό και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το χρονοδιάγραμμα από πλευράς μας. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και με ικανοποιεί ότι μπορούμε να διεξαγάγουμε αυτή τη σημαντική ε, μεγάλη εμβέλεια συζήτηση σήμερα και να μπορέσουμε να δούμε τα θέματα των πέντε αυτών κρατών και να δούμε από πλευράς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι μπορεί να γίνει με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναμείνουμε ώστε να υπάρξουν τα νέα στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν ίσως τη δυνατότητα να επανατοποθετηθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Helmut Σόλτς. Και τώρα, σε σχέση με την έκθεση που μας δώσατε, έχω την τιμή και την χαρά, μια και έχουμε τον Υπουργό Εμπορίου της Κένιας ανάμεσά μας, να μπορέσω να του δώσω τον λόγο να παρέμβει. Να μας αποσαφηνίσει κάποια πράγματα για αυτές τις διαδικασίες. Και φυσικά θα μας περιγράψει και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα για την Κένια. Παρακαλώ, και τον λόγο. Very Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Εκ μέρου ε, της κυβέρνηση και του λαού της Κένιας ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας ε, δίνει τη δυνατότητα να ε, απευθύνουμε το λόγο σε εσά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κένιας ε, για το, μέχρι το 2018 που ξεκίνησε το 2007 για μένα, ε, καθώς και για τους ε, κυβέρνηση και για τους ιδιώτες εταίρους που επηρεάζονται φυσικά από αυτή τη συμφωνία, και ε, έχουμε εδώ και τον ε, πρέσβη μας. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαρήκαμε που σας συναντήσαμε όταν στα πλαίσια, στο περιθώριο της συνάντησής μας αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τα 40 χρόνια και πλέον ε, αφορολόγητης πρόσβασης που είχε παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κένια μεταξύ άλλων πρωτοβουλειών αναπτυξιακών που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει το λαό της Κένιας. Οι προτιμησιακές ε, δασμολογικές ε, καταστάσεις οι οποίες ε, μας προσφέρατε, μας επέτρεψαν να έχουμε πρόσβαση σε μια φορολόγητη αγορά και μπορούσαμε να έχουμε εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι η αγορά εξαγωγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, ε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη είναι φαινόμενο όπως ε, φαίνεται από τα εξής. Πρώτον, έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους, ε, οι, κυρίως ε, γυναίκες και νέους, κυρίως στις περιοχές της Υπέθρου, που βγάζουν τα προστοζήν είτε άμεσα είτε έμεσα από επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ε, τεράστιες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες ανέρχονται σε πάνω από 2 δις ευρώ, ε, και ε, γίνονται για επιχειρήσεις οι οποίες ε, παράγουν αποκλειστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, τεχνογνωσία που επέτρεψε στους γεωργούς στην Κένια να αναπτύξουν τη γεωργία και να έχουμε ωφέλη και για τη χώρα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχουμε βοήθεια ε, στους καταναλωτές, κυρίως ε, τους καταναλωτές που αγοράζουν ε, λουλούδια από την Κίνα και ε, αυτό έχει βοηθήσει ε, λόγω των προτιμησιακών δασμών που προσφέρονται στη γηγένεια. Οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί σε ισχυρή ε, ολοκλήρωση η οποία έχει βοηθήσει χάρη και στους κανόνες καταγωγής. Υπάρχει μεγάλη ε, ανάγκη και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρωτοβουλία της περιφερειακής ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει και την Τελωνιακή Ένωση καθώς επίσης και την Κοινή Αγορά και την Νομισματική Ένωση. Ε, είναι ο κύριος προορισμός των εξαγωγών της Κίνας ε, η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίση έχουμε και πολλά ωφέλη από χώρες εταίρους ε, της κοινή αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για μας ως χώρα. Κύριε Πρόεδρε, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ένας στόχος ε, και της Κένιας και οι εταίροι μας χρησιμοποιούν με άλλες ε, περιοχές, όπως επίσης ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΕΝΤΑΚ ε, και άλλες. Θέλουμε να ενισχύσουμε την περιοχή και να είναι προορισμός και χώρος προέλευσης προϊόντων προς εξαγωγή όσον αφορά την ευρύτερη ολοκλήρωση. Οι διάφορες ε, αρχές μας ε, υπάρχουν ε, και συμμετρικά αλλά και με ασυμμετρία. Έτσι μπορέσαμε να τηρήσουμε κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μεταξύ μας αλλά και με άλλες ε, ομάδες ε, εμπορικών συμφερόντων και φυσικά αυτό είναι προσόφελος όφελος ε, των οικονομιών της περιοχής χωρίς να ζημιώνουμε το στόχο της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Όσον αφορά τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, από το 2007 ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2014. Η συμφωνία αυτή θεωρείται από την Κένια και άλλες ε, χώρες ε, της Ανατολικής ε, Αφρικής ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Η απόφαση να την υπογράψουν όλες οι χώρες εταίροι έχει ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών των χωρών της Ανατολικής Αφρικής και επικυρώθηκε και από τη Σύνοδο Κορυφής που έγινε ε, το Μάρτιο του 2016. Ε, η ε, επόμενη φάση είναι να υπάρξει μια ημερομηνία στην οποία θα υπογράψουν όλες οι χώρες για να προχωρήσουμε ε, και να συστήσουμε επίσης και ένα τεμεακό συμβούλιο για τις χώρες ε, αυτές ε, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η υπογραφή της συμφωνίας στις 18 Ιουλίου όμως δεν έγινε όπως είπατε κύριε Πρόεδρε διότι υπήρχαν κάποιες εξελίξεις στην περιοχή και περιφερειακά αλλά και διεθνώς. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μία σύνοδος ε, κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να μπορέσει να συζητηθεί το θέμα της υπογραφής της συμφωνίας από κάποια από τα κράτη-μέλη. Λόγω της ε, μοναδικής θέσης της Κένιας όμως, από τον Ιούλιο του 2016, έχουμε δεσμευτεί και με τις χώρες εταίρους μας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα υπογράψουν τη συμφωνία όπως είχαμε συμφωνήσει αρχικώς. Έγιναν αρκετές ε, συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών, ε, ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και να ολοκληρωθεί επιτέλους. Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η Σύνοδος Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια κατεύθυνση για το τι ακριβώς θα κάνουμε οι διαδικασίες καθώς επίσης και η συνθήκη ε, δεν ε, παρακολύονται όμως. Τίποτα δεν απαγορεύει σε καμία χώρα να ε, υπογράψει τη συμφωνία γιατί έχει ήδη ληφθεί απόφαση προηγουμένως. Το σενάριο είναι αντίστοιχο με τον Οκτώβριο του 2014 που είχαμε τη μονογραφή της συμφωνίας στις Βρυξέλλες και αυτό οδήγησε φυσικά την μονογραφία από τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν διατεθειμένα να μονογράψουν και επιτρέπεται και ε, στα κράτη-μέλη που δεν είναι ακόμα έτοιμα να ε, συνεχίσουν τις διαβολεύσεις και να συμμετέχουν αργότερα αν το επιθυμούν. Τα πέντε κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να υπογράψουν, κύριε Πρόεδρε, αμέσως τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα υπόλοιπα κράτη, όταν θα είναι έτοιμα, ε, θα συμμετέχουν και αυτά και θα υπογράψουν την συμφωνία εν ευθέτω χρόνο. Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα. Όπως γνωρίζετε, ε, η πρόσβαση της Κένιας από το 2014 σε μη δασμολογικούς ε, φραγμούς ε, έχει την υποχρέωση να κυρώσει την τη συμφωνία μέχρι το 2014. Η Κένια ε, χαίρει και της ε, κατεξουσιοδότησης πράξης, ε, ε η οποία ε, χρησιμοποιείται σε περίπτωση που η Κένια δεν μπορέσει να υπογράψει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Ε, δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει μετά το 2016 μέχρι την 1η Οκτωβρίου που λύγει η προθεσμία. Εάν ε, ε άρετε την πράξη εξουσιοδότηση θα υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Η χώρα θα χάσει το δεύτερο πιο σημαντικό προορισμό ε, εξαγωγών της ε, εν μία νυχτή. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει τεράστια πόλια θέσεων εργασίας που θα επηρεάσει πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους στην γένεια. Επίσης μπορεί να κλείσουν και πάνω από 200 επιχειρήσεις και να χαθούν επενδύσεις άνω των 2 δις ευρώ. Και φυσικά αυτό ε, θα δημιουργήσει και προβλήματα αστάθειας, ε, ανεργίας, ε, κυρίως μεταξύ των νέων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται στις εκμεταλλεύσεις οι οποίες εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και ένας μεγαλύτερος πονοκέφαλος διεθνώς, διότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κοιτάξουν σε άλλες περιοχές αλλού θα δημιουργήσουν ε, και περαιτέρω κύματα μετανάστευσης που, ανθρώπων που θα στραφούν σε άλλες χώρες του κόσμου και φυσικά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, φυσικά θα επηρεάσουν και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Ανατολικής Αφρικής. Υπάρχουν ε, ε, σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών και των επιχειρήσεών τους. Επομένως η Κένια θα ήθελα να ζητήσει από την Επιτροπή σας να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να διασφαλίσετε ότι η πρόσβαση στην αγορά που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή η Κένια δεν θα τύχει προβλημάτων και ότι αυτό θα είναι εις βάρος και τη Κένιας αλλά και τη περιφερειακή οικονομία θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά βάσει της συμφωνίας, αυτό θα γίνει για όλες τις υπόλοιπες χώρες εκτός από την Κένια. Για να ε, προλάβουμε τέτοιες απώλειες, ε, επειδή ακριβώς δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, θέλουμε να φροντίσουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία ως περιοχή. Επίσης, έχουμε εγκρίνει τα εξή μέτρα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει των ε, συγκεκριμένων συνθήκων. Πρώτον, έχουμε γράψει επίσημη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να υπογράψουμε τη συμφωνία αμέσω ω Κένια. Επίσης είπαμε ε, ότι τουλάχιστον δύο από τις πέντε χώρες έχουν δεσμευθεί να υπογράψουν τη συμφωνία αμέσως μαζί με εμάς. Κάποιες άλλες έχουν υποδείξει ότι σκοπεύουν να την υπογράψουν μετά από τη Σύνοδο Κορυφής που προβλέπεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά την υπογραφή, η Κένια δεσμεύεται να ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης και να περάσει από το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, έχουμε ζητήσει μια έκτακτη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία έχει προγραμματιστεί προς το παρόν προσωρινά για τις 8 Σεπτεμβρίου, ε, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε και την υπογραφή των υπολείπων ε, χωρών μελών και ε, κυρίως ζητάμε να λάβετε γνώση της συνεχούς δέσμευσης της Κένιας ε, για να εμβαθύνουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση και φυσικά ε, και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, να λάβετε γνώση και της απόφασης της Κένιας και τουλάχιστον ενός άλλου μέλους να υπογράψει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία. Δεύτερον, θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει καμία διακοπή στο σύστημα ε, φορολόγησης ε, των προϊόντων, ε, των αφορολόγητων προϊόντων και ελπίζουμε ε, να λάβετε υπόψη και το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από την έκτακτη Σύνοδο κορυφή το Σεπτέμβριο. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, ε, σημειώνω με χαρά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η Γένεια από Οκτωβρίου θα έχει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέχρι να υπογράψει και να κυρώσει τη Συμφωνία η και εμεί θέλουμε να την υπογράψουμε και να την κυρώσουμε. Επίσης, ε, θεωρούμε, όπω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτή δεν είναι η βέλτιστη δυνατή λύση και θα προσπαθήσουμε να υπογράψουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Όμως, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των ε, μελών υπογράψει και εμεί θα το επιδιώξουμε αυτό και η Κένια θα κυρώσει τη συμφωνία, η Κένια θα ήθελε να διατηρήσει την πρόσβαση στην αγορά βάσει της συμφωνίας ε, και όχι βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για το σαφές αυτό μήνυμα που μας ε, στείλατε. Οι σκιώδεις εισηγητές ε, τώρα, παρακαλώ, το ΕΛΚ, κύριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρίως εγκρίνω την άποψη του εισηγητή του κυρίου Χέρμουτ Σόλτς όπως ε, μας την εξέθεσε. Και σας ευχαριστώ κύριε Σόλτς για την παρουσίασή σας, για την έκθεσή σας. Πολύ συνθετική αλλά και πολύ περιεκτική και παρουσιάσατε το συνολικό πρόβλημα το οποίο ιστορικά μας παρακολουθεί μέχρι σήμερα και κατανοώ ότι από πλευράς του εισηγητού το κείμενο αυτό πρέπει ακόμα να αναμένει την τελική παρουσίασή του διότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα ακόμα. Τα αφρικανικά κράτη, το σύνολο ίσως και όλα της Αφρικής είναι μια πάρα πολύ σημαντική ε, περιφέρεια, μια πάρα πολύ σημαντική ενότητα και όχι μόνο για οικονομικούς ή εμπορικούς λόγους που πάντα υφίστανται αλλά και είναι πάντα η βάση για τέτοιου είδους συμφωνίες αλλά και για πολιτικά ζητήματα. Πρόκειται ακριβώς και για κοινωνικά ζητήματα και τα τελευταία χρόνια έχουμε και γεωπολιτικά ζητήματα όπως θα έπρεπε να τα αποκαλέσουμε για τους πιο διαφορετικούς λόγους που επηρεάζουν τα πράγματα και που για παράδειγμα με την Ανατολικοαφρικανική κοινότητα αλλά και με τις άλλες συμφωνίες ε, δημιουργούν κάποια ζητήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία και εδώ προστίθεται και ένα άλλο επιπρόσθετο ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται και το ανέφερε ο κύριος εισηγητής. Δηλαδή η προσέγγιση από πλευράς της, των κυβερνήσεων σε σχέση με τις διάφορες χώρες των αφρικανικών, των, της κοινότητας των αφρικανικών χωρών εδώ δεν είναι μόνο θέματα εκπροσώπησης κρατών και συμφερόντων τους, αλλά και θέματα κομματικά τα οποία αφορούν μια κυβέρνηση και τα οποία παρισφρέουν και είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσουν σε μια διευθέτηση των θεμάτων, διότι δημιουργείται μια πολύ ε, δυσχερής κατάσταση, είναι μια πολύ σημαντική κατάσταση, για παράδειγμα στην Ανατολική Αφρική, η Κένια. Και αυτές οι δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από την άλλη πλευρά όμως έχουμε χώρες ε, όπως την Τανζανία και υπάρχουν προβλήματα εκεί με την ίδια την δυνατότητα λήψης απόφασης από πλευρά τους ή κατάληξης σε μια συμφωνία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και εμείς αυτά τα θέματα στα θέματα τα οποία θα πρέπει να σταθμίσουμε για να λάβουμε μια απόφαση και να γνωρίζουμε και τις απόψεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε μια και πρόκειται για σημαντικά θέματα θα πρέπει δεν χρειάζεται εδώ να επαναλάβουμε όλα τα στοιχεία αλλά πρόκειται για την κατεύθυνση και την διαμόρφωση της γνωμοδότησης όχι μόνο εγώ αλλά όλο το κόμμα μας θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι σημαντική και οι άλλες συμφωνίες επίσης είναι σημαντικές και πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ολοκλήρωση με συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία θα αφορούν ε, τις χώρες αυτές που πρέπει να τύχουν τις συνδρομή μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τον πιο εύθετο τρόπο και χρειάζεται εδώ μια αναβαθμισμένη προσπάθεια αλλά και νυφαλιότητα και σύνεση που πρέπει να πριτανεύει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και συνολικά. Και συμφωνώ με την άποψή σας ότι με την έναρξη σε ισχύ αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να ολοκληρωθεί το δυνατόν ταχύτερα για να αρχίσει να ισχύει. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα θέματα προθεσμίας τα οποία δημιουργούν και αυτά από πλευρά τους κάποιες δυσκολίες. Θα πρέπει να ζητηθεί λοιπόν να παρουσιαστούν οι θέσεις των διαφόρων εταίρων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε διότι από την άλλη πλευρά επιθυμούμε πράγματι να αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία. Αφετέρου όμως έχουμε διαφορετικούς εταίρους απέναντί μας, όπως για παράδειγμα την Κένια, με ιδιομορφίες που ε, χαρακτηρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αντιμετωπίζουν και προβλήματα σε σχέση με συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε συγκεκριμένη κατάσταση σήμερα. Από την άλλη πλευρά έχουμε για παράδειγμα το Μπουρούντι και πάλι τέτοιου είδους χώρες έχουν προβλήματα ξεχωριστά με την υπογραφή αυτών των συμφωνιών. Περί τίνος πρόκειται ε, για αυτά τα προβλήματα για αυτές τις χώρες. Πρόκειται για την ρήτρα εκπνοής, ε, την ρήτρα κατάληξης. Και πρέπει εδώ να δούμε το ευτυχές γεγονός μέσα σε μια ατυχία ή σε μια ε, κατάσταση και να δούμε πώς είναι δυνατόν να ε, αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά των χωρών αυτών και για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ελευθεριών που πρέπει να διασφαλίζονται υπέρ των πολιτών αυτών των χωρών. Και πρέπει να δούμε ότι κατά την προηγούμενη ε, κατά το παρελθόν ήταν το πιο επιτυχές μέσο αυτό για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε αυτές τις χώρες ώστε να σέβονται και να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οικονομικά μέσα λοιπόν και συμφωνίες που θα πρέπει βοηθώντας, συνδράμοντας τα κράτη αυτά να διασφαλίζουν από την άλλη πλευρά την τήρηση αυτών των αρχών. Αναμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθούν διαδικασίες και να κατατεθεί η γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε πολύ και έχετε τώρα εσείς τον λόγο. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό για τα όσα μας είπε. Και τον Χέλμουτ βέβαια για την μακρά εισαγωγή που μας έκανε όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή, και τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας. Το πρώτο, η πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι να υπάρχει συνοχή αναπτυξιακής πολιτικής και εμπορικής μας πολιτικής όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών οικονομικής εταιρική σχέσης. Είναι σαφές ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη σε κάθε μία από τις χώρες. η απόφαση της Τανζανίας για αναβολή της υπογραφής της συμφωνίας καταδεικνύει ότι υπάρχουν ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουνα υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα με, την, με το αποτέλεσμα κινδυνεύει να υπάρξει κάποια ανισορροπία. Υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την ε, βιομηχανία και άλλες πολιτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα, για τον Μπουρούντι. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους, που πραγματικά δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία το Μπουρούντι και εφόσον ανεργοποιήθηκε το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού, ε, θέτει που αμφισβήτηση όλες τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι ισορροπία υπάρχει σε αυτήν τη συμφωνία. Έγιναν πολλά σχόλια για τα οικονομικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας αυτής και τα δοσμολογικά της χαρακτηριστικά. Αλλά από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχοντας ακούσει για τις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες τέτοιες συμφωνίες, διαπιστώνουμε ότι εδώ δεν υπάρχει αρκετή εξασφάλιση. Κυρίως στον Μπουρούντι. Η κατάσταση είναι τέτοια που μας αναγκάζει να ξαναδούμε τη διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες μας. Αν θέλουμε να υπάρχει συνοχή και να προβλέπεται ανάπτυξη. Δεν υπάρχει κεφάλαιο ε, παρκές για την αηφόρο ανάπτυξη. Είναι κάτω από τα όρια που έχει θέσει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις οικονομικές της συμφωνίες. Και σίγουρα είναι κάτω από τα όσα συμφωνήσαμε εμείς σε άλλες οικονομικές συμφωνίες με Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μη τι άλλο, να είχε κάνει κάτι για τις σχέσεις μας με την κοινότητα των χωρών Ανατολικής Αφρικής. Όμως δεν το κάνει. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ενοχλούμε και βάζουμε σε δύσκολη θέση τη μόνη χώρα η οποία ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει περισσότερο. Συστήσαμε για τις κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά τώρα για την Κένια, με τη κατεξουσιοδότηση πράξης θα έβγαινε η Κένια από τις χώρες με τις οποίες θέλαμε να προχωρήσουμε. Ενώ στόχος είπαμε ότι είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση και συμφωνίε ε, περιοχής με περιοχή. Πρέπει όμως να είναι και οι χώρες εταίροι μας μέσα. Αλλιώς πάμε πίσω στις σκοτεινές περιόδους ε, διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση. Και ακούσαμε τους συναδαρφούς με τις διάφορες ιδέες τους Πολλές ιδέες ακούγονται όντως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από πλευρά τη κυβέρνηση τη Κένια. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση για την Κένια, ώστε να υπάρχει πρόσβαση χωρί δασμού και χωρί ποσοστώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ζητάω να έρθει με λύση. Και ενώ έχουν αναβάλει την υπογραφή οι χώρες, εγώ ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της συμφωνίας. Να κοιτάξει πώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες της περιοχής, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει το Brexit σε τέτοιου είδους συμφωνίες, τι σημαίνει για την ισορροπία των συμφωνιών. Να βελτιώσουμε επίσης τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και τα σχετικά κεφάλαια και να φροντίσουμε να υπάρχει εποπτεία από την κοινωνία των πολιτών και από μικτές κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Είναι ζωτική συμφωνία, αν θέλουμε μια συμφωνία που να προωθεί και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη. Χωρί αυτά τα στοιχεία, οι συμφωνίε μα θα είναι συμφωνίε πρώτη γενιά, εμπορικέ και όχι δεύτερη γενιά. Εμείς περιμένουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ σε ευχαριστούμε. Για τον κύριο Κέμπελ, ποιος τον αντικαθιστά, ο κύριο Στάκουλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ναι, τον αντικαθιστώ. Αντικαθιστώ την κυρία Σάρκερ, μάλλον. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τις, τη συμφωνία αυτή οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες τη κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής πρέπει να πετύχουν οι συμφωνίες. Όπως ξέρετε, δεν πρόκειται για μια κλασική συμφωνία μπορική, αλλά πρόκειται για μια συμφωνία προοδευτικού χαρακτήρα, σημαντική και για την ανάπτυξη. Εμείς, οι ευρωβουλευτές, πρέπει να ζητάμε να εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες. Έπειτα, όσον αφορά την διαδικασία κύρωσης, Πρέπει να βγούμε από τα διέξοδο οπωσδήποτε και να βρούμε μια λύση για την Κένια. Η συμφωνία πρώτα απ' όλα είναι σταδιακή και ασυμμετρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει πλήρως τις αγορές της στις χώρες ΑΚΕ, ενώ εν μέρη και με προσωρινές περιόδους. Ωραία, σαν σημείο κίνησης είναι καλό αυτό. Όμως θα ήταν καλό να υπάρξει και εποπτεία και άνοιγμα της αφρικανικής αγοράς σε επίπεδα τα οποία να είναι ικανοποιητικά και με περιόδους προσαρμογής που να επιτρέπουν στις χώρες να προσαρμοστούν. Είναι ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία ε, θα είναι υποφελής για όλες τις οικονομίες. Δεύτερον, η Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση πρέπει να ευνοεί την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Ανατολική Αφρική. Είναι ζωτική σημασία στο βαθμό που οι Αφρικανοί εταίροι μα εργάζονται προκειμένου να υπάρξει μία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στην Ήπειρό τους και πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε για αυτή την ολοκλήρωση. Τρίτον, οι συμφωνίες αυτές πρέπει οικονομικά και κοινωνικά να αποτελούν εργαλεία για την ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι ρήτρε για πέντε χρόνια να ανανεώνονται ανάλογα με τις εξελίξεις. Βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης. Η απλή μνήα τη Συμφωνίας σκοτονού, δεν φτάνει. Οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αρκετά ισχυρές κατά τη γνώμη μου. Τέλος, η συμφωνία αυτή έχει βρεθεί σε ένα στάδιο που δεν προχωράει πια, λόγω της Κένιας. Τώρα θα έπρεπε να προχωρήσουμε με περισσότερη φιλοδοξία δεδομένου η Τανζανία και η Ουγγάντα έχουν προχωρήσει περισσότερο. Πρέπει να βρεθεί και μια εναλλακτική λύση, αν τελικά οι διάφορες πλευρές αρνηθούν να υπογράψουν. Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε την Κένια να υποφέρει εξαιτία μια κατάσταση για την οποία η χώρα ίδια δεν έχει καμία ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Λούνς, εσείς, όχι, η κυρία Σκά Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν, οπότε θα φροντίσω να είμαι σύντομη. Σίγουρα δεν έχει νόημα να έχουμε τώρα εξουδιώτηση πράξη για την Κένια. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν δεν θα την αποσύρει. Να μας πει τέλο πάντων, για να είναι ξεκάθαρο για μας, τι θα κάνει. Αν η Τανζανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τι συνέπειες από το Brexit, νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Στο κατω όλοι θα θέλαμε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες θα είναι επιπτώσεις από το Brexit. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι αρκετή δικαιολογία, ότι δεν είναι σωστό ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να ζητήσει κανείς ε, παράταση. Και πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης. Το Συμβούλιο πρέπει να κυρώσει το κείμενο, αν το πήρε πάνω από ένα χρόνο, έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε σε διαδικασία επιταχυμένη. Οπότε γιατί να πετήσουμε κάτι τέτοιο από άλλες χώρες, να είναι πιο γρήγορες από μας. Οπότε συμφωνώ με τις επικρίσεις για τη στάση αυτή. Τώρα, συνάδελφοι, και για την Κένια έχουμε δει και άλλη φορά τις συνέπειες. Οπότε αυτή τη φορά προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η Τζουντ για τη συμφωνία αυτή, αλλά είναι πράγματι σημαντικό να μιλήσουμε για τις συμφωνίες μιας νέας γενιάς για την Αφρική και να δούμε τις νέες δεσμεύσεις του ΟΗΕ όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και όσον αφορά το COP21. Σήμερα, στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών, δεν το συζητάμε καθόλου. Κρίμα, γιατί οι διαπραγματεύσεις βέβαια είναι ετών πια τώρα. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να μπορέσουμε τα νέα δεδομένα να τα συμπεριλάβουμε στις νέες σχέσεις που έχουμε με τις αφρικανικές χώρες και στις εμπορικές μας σχέσεις μαζί τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε μετά το κοτονού τι γιατί ξέρουμε ότι οι εμπορικέ συμφωνίε ενσωματώνονται στη Συμφωνία Κοτονού που λήγουν το 2020. Έχουμε σαν σημείο αναφορά σε αυτές τις συμφωνίες Κοτονού, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο η ισχύση ή μη ισχύση του Κοτονού κάνει και αυτές τις συμφωνίε να ισχύουν ή όχι, ανάλογα. Δεν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση επίσης για την ε, δέσμευση απέναντι στο Κοτονού. Και υπάρχει και το θέμα της ε, δεσμευτικής ε, στάσης απέναντι σε διάφορα σημεία της συμφωνίας. Δουλεύουμε για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αφρική για να συνάδουμε με τον ΠΟΕ. Αυτό ακούμε πάντα. Αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό να είμαστε δηλαδή εντάξει με τις διατάξεις του ΠΟΕ. Θα ήταν λοιπόν πιο χρήσιμο να δουλεύουμε κυρίως για να μην πω αποκλειστικά σε αυτή τη συμμόρφωση, αντί να ε, ε, κάνουμε χώρες όπως οι τέσσερις στις πέντε που είναι χώρες EMA που ε, βρίσκονται προβλήματα ανάπτυξης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα γιατί υπάρχει απελευθέρωση 82% ενώ η Ευρώπη 90%. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου οι χώρες αυτές όπως η Ουγγάντα και η Τανζανία, το Μπουρούντι, η Ρουάντα βρίσκονται σε κατάσταση ανάπτυξη που είναι πολύ πιο κάτω από το δικό μας επίπεδο ανάπτυξης στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λοιπόν μηχανισμός προστασίας για αυτούς. Και τώρα θα επανέλθω με πολιτικά σε αυτό που είπα και πριν, ότι η Ευρώπη ε, πρέπει να μην υπογράψει εύκολα συμφωνία με τον Μπουρούντι. Το Ιούλιο του 2016 είχαμε μια έκθεση από τον ΟΗΕ που αναφέρεται στον Μπουρούντι και λέει 342 εκτελέσεις μέσα σε ένα χρόνο. Εκτελέσεις συνοπτικές, 200 ε, περίπου πολίτες που βρέθηκαν επίσης σε κοινούς τάφους γύρω από την Μπουζουμπούρα. Εμεί λοιπόν τι κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία με μια κυβέρνηση που είναι τέτοιου είδου κυβέρνηση στην Ανατολική Αφρική. Ρωτάω λοιπόν, όπω ρώτησε και ο υπουργό τη Κένια, θα γινόταν να έχουμε συμφωνία η οποία να αφορά δύο ή τρεις χώρες από αυτή την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας είχε πει όχι. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με πέντε χώρε και συνεπώσει η ευρωπαικη επιτροπη αρχικα μας ειχε πει οχι οι διαπραγματευσει εγιναν με πεντε χωρε και συνεπω η συμφωνια θα αφορά και τι πέντε. Ε, ρωτάω, η συμφωνία αυτή μπορεί να γίνει μόνο με μία, δύο χώρες που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Έτσι, λύνεται το ζήτημα της Κένια σε σχέση με τις άλλες χώρες οι οποίες αρνούνται να υπογράψουν, αλλά λύνει και το δικό μας ευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν θέλουμε να υπογράψουμε μια συμφωνία με τον Μπουρούντι. Άρα παραμένει το ερώτημα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα σχέδιο Β που θα ήταν το GSP συν. Πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ότι είναι εναλλακτική στο GSP, αλλά ποτέ δεν μίλησε για το GSP συν. Θα ήταν ίσω και για την Κένια μια ενδιαφέρουσα λύση, γιατί θα επέτρεπε στην Κένια να μην σπάσει με τη λογική τη περιφερειακή ολοκλήρωση, γιατί δεν θα ήταν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ευρώπη Κένια, αλλά θα ήταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε στην Κένια να έχει πρόσβαση στι ευρωπαϊκέ αγορέ χωρί όμως να δυσκολεύει τις άλλες τέσσερις χώρες. Η εναλλακτική αυτή λύση έχει εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου η Κένια να μην βρεθεί σε μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε αστάθεια την οικονομία της. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω για ένα-δυο λεπτά που το προτιμώ από το να συμμετείχα στην όλη διαδικασία γιατί είναι τόσο περίπλοκη. Ε, έχουμε τις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης, ε, το ΜΑΡ, το Κοτονού, να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να με εξηγήσετε όμως κάτι, διότι αυτή η συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί, εγώ έφτασα βέβαια τώρα, αλλά είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Τη συζήτηση για την εκπνοή αυτού του κανονισμού. Γνωρίζουμε ότι ο λόγος είναι ότι κάποιες χώρες δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει τις ε, συμφωνίες, αλλά με χαρά ακούω ότι η Κένια δεσμεύεται να υπογράψει και να κυρώσει τη συμφωνία, τουλάχιστον από πλευρά τη. Και αν το κάνουν, ε, λογικά το πρόβλημα θα πρέπει να θεωρείται λήξαν. Διότι η πράξη κατεξουσιοδότηση λέει ότι θα διατηρήσουν την προτιμησιακή πρόσβεση Ω συνέπεια αυτού ε, αν έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία. Και αν πιστέψουμε αυτό που ακούμε, και εγώ το πιστεύω, τότε εγώ δεν μπορώ να δω που βρίσκεται το πρόβλημα και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Και βεβαίω θα μπορούσε κανείς να αντιστρέψει το όλο ζήτημα και να πει ότι είναι αυτό κάποιο καινούριο πρόβλημα. Θα ήθελα να ακούσω τη δέσμευση της Κένιας, αλλά με εκπλήσει λίγο το γεγονός ότι γίνεται τώρα η συζήτηση. Το παραπέντε. Θα μπορούσαμε βέβαια να συζητούμε αν είμαστε στο και πέντε πλέον ε, για το θέμα της κύρωσης υπογραφής. Θα έπρεπε να είχε γίνει η συζήτηση πριν από δύο μήνες, γιατί δεν θα βρισκόμασταν ενώπιον αυτής της κατάστασης τώρα. Ακούω ότι κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά θα ήθελαν μια καθυστέρηση. Εγώ δεν είμαι εξ αυτών που είναι υπέρ της καθυστέρησης και ο λόγος είναι ότι Όσα χρόνια είμαι εδώ, ε, πάντα ακούμε το θέμα αυτών των συμφωνιών. Έχει καθυστερήσει περισσότερο από όλα, έχει πάρει πολύ περισσότερο. Δεν είχαμε μόνο σχέδιο Β, σχέδιο Γ, ενδιάμεσες συμφωνίες. Προσπαθήσαμε με διάφορες ιδέες και τρόπους να ε, κινήσουμε το ζήτημα. Και υπ' αυτή την έννοια, πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή πρόταση της Μαρία Ρένα να δούμε το GSPC αλλά από πλευράς ε, της Κένιας ε, θα πρέπει να υπάρχει, να, να κάνουν τι, να κάνουν αίτηση και μετά να κυρώσουν τις 27 συμβάσεις. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή, αλλά πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα αυτή η ιδέα με την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνίας. Γιατί άπαξ και γίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα. Τουλάχιστον όχι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και μετά θα πρέπει να καταλάβουμε... ένα σαφές ε, μήνυμα προς ε, τους προσκεκλημένους μας. Τι θα γίνει αν έχει επικυρώσει την ε, Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Λύνεται τότε το πρόβλημα και έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς δασμούς, ποσοστώσεις κτλ. Μπορείτε να μας το αυτό και να απαντήσετε και σε υπόλοιπε ερωτήσεις των συναδέρφων. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Υπουργό που ήρθε εδώ και μας παρουσίασε την επιθυμία της χώρας του να παραμείνει μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δέσμευση, γιατί και εμείς προσβλέπουμε να επεκτείνουμε μάλιστα και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε όλες τους όχι μόνο το εμπόριο. Γνωρίζουμε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα αρχίσω λοιπόν τονίζοντας ότι παραμένει ο βασικός μας στόχος που είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση. Νομικά μιλώντας, οι χώρες ΑΚΕ έχουν δεσμευτεί στη διάσκεψη ήδη να υπογράψουν, μάλλον στις συνεδρίες των Υπουργών ε, Εμπορίου. Οπότε όλε οι χώρες είναι ελεύθερε να υπογράψουν τώρα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο, μπορούν να υπογράψουν, θα υπογράψουν, οπότε νομικά μιλώντας προχωράμε. Αν υπογράψει και κυρώσει η Κέννη, όπω είπε και νωρίτερα, δεν είναι ότι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία εταιρική σχέση, αλλά ότι θα παραμείνει η Κένια όπως ήταν, αυτό σας είπαμε. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδίας τον κύριο Σόλτς, γιατί πραγματικά ετοίμασε κάτι πάρα πολύ αντικειμενικό και έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση μιας συμφωνίας που σίγουρα είναι περίπλοκη όπως είναι και όλες αυτές οι εταιρικέ σχέσεις. Σίγουρα χρειάζεται να καταλάβει κανείς και του είμαι ευγνώμων που ανέφερε και τις επιθυμίες για την βιώσιμη ε, ανάπτυξη, μη εκτέλεσης κλπ. κλπ. Πρόκειται για μια ε, συμφωνία η οποία σίγουρα κυστρώνεται στη Συμφωνία Κοτονού. Και είμαι επεπισμένη, όπως ήμουνα και πριν, ότι πρόκειται για μια ρήτρα η οποία δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι δυνατότητες που θέλει να έχει. Δηλαδή να εξετάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Τώρα, να μην υπάρχει αμφιβονία ούτε εγώ ούτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μιλάμε για το GSP αντί για το GSP συν. Το GSP είναι αυτό το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε χωρίς να συμβεί τίποτα άλλο. Ενώ το GSP συν πρέπει να υπάρξει αίτηση για να προχωρήσουμε σε αυτό. Οπότε δεν είναι αυτή η λύση για να διατηρήσουμε τα προνόμια εφόσον δεν υπάρξει ε, συμφωνία εταιρική σχέσης. Τώρα η χώρα σαφώς και θέλει ε, βάση θυσία και προτιμάει μια συμφωνία εταιρική σχέσης αντί για GSP ή GSP συν. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που αναφερόμουν στο GSP και όχι στο GSP συν. Τώρα, είναι μια συμφωνία αυτή με μια περιφέρεια με μεγάλη ελευθέρωση. Τα 5% του εμπορίου της είναι ήδη σε μηδέν όσον αφορά το MFM, δηλαδή τους, με τους εταίρους του ΠΟΕ. 17% όσον αφορά τον όγκο εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι διαχειρίσιμο, γιατί η περιοχή αυτή έχει ένα μορατόριο με 7 με 12 χρόνια, συν 25 χρόνια εφαρμογή. Άρα μιλάμε για το 2023 ως τελευταίο έτος εφαρμογής. Δεν νομίζω ότι είναι διχειρήσιμο αυτό για το 17% που πρέπει να ελευθερωθεί από πλευρά Ευρώπη. Βάλτε δίπλα και το κεφάλαιο για την αναπτυξιακή συνεργασία, που είναι ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκε περισσότερο με τη ρήτρα μη εκτέλεση. Το κεφάλαιο αυτό λοιπόν είναι ζωτική ε, σημασία γιατί είναι μια περιφέρεια που χρειάζεται τις υποδομές για να μπορέσει να συνεχίσει την τάση της να αποτελεί ένα ε, λιμένα στην ε, Αφρική, ένα λιμένα προστασίας εντό εισαγωγικών, hub, ένα κόμβο. Δεν ε, θα μπορούσα πάντως παρά να συμφωνήσω με αυτά που είπε και η κυρία Κιπάλανα, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνοχή για την ανάπτυξη. Και γι' αυτό και εμείς θέλουμε μια περιφερειακή συμφωνία και είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε, ιδιαίτερα μετά από αυτά που μας είπε ο αξιότιμος υπουργό της Κένια σήμερα το πρωί. Τέλος. για να απαντήσουμε στο πώς μπορούμε να αποφύγουμε την καταστροφή για την Κένια, ε, αυτό θα γίνει αν παραμείνει η Κένια στο ΜΑΡ. Αλλά αν έχουμε όλες τις υπογραφές και τις κυρώσεις, τότε θα έχουμε την ε, Οικονομική Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουτ, παρακαλώ. Κύριο Ερώτηση ήταν, ε. κατάλαβα καλά, εάν η Κένια υπογράψει και κυρώσει, τότε βάσει της πράξης εξουσιοδότηση, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι, δηλαδή αν κάνουν αυτό που μας πούμε, τότε δεν υπάρχει, που μας είπαν ότι θα κάνουν, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, βάσει της ε, ΜΑΡ. Ο Ντανίλ Κασπαρή για να το διευκρινίσουμε, γιατί έγινε και αυτή η συζήτηση και το πρωί και πάλι. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν κάποια μέλη για την Κένια, με βάση αυτή την πράξη κατεξουσιοδότηση, ε, ε Ναι, η πράξη κατεξουσιοδότηση καλύπτει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Καταρτήσαμε τις πράξεις εξουσιοδότηση με βάση τις διάφορες περιπτώσεις και για την Κένια είναι σαφές ότι η κύρωση της συμφωνίας του 2014 τους δίνει τη δυνατότητα να μείνουν στη ΜΑΡ. Ε, τονίζω τη ΜΑΡ που σημαίνει ότι δεν είναι όπως η ενδιάμεσα συμφωνία της ακτής του Ελεφαντιστούν ή της Γκάνα που είναι ένα ισχυρό μέσο το οποίο είναι συμβατό και με τον ΠΟΕ. Η ΜΑΡ είναι τελείως διαφορετικό μέσο. Η κυρία Ρένα, για να είμαι βέβαιη, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτό σημαίνει υπογράφουμε, κυρώνουμε, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η συμφωνία δεν ε, θα εφαρμοστεί γιατί τα άλλα τέσσερα μέλη δεν υπογράφουν. Αυτά τους δίνει πρόσβαση στην αγορά και ε, έχετε μια συμφωνία για τον ΠΟΕ, για μια συμφωνία που ξέρετε ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Αν είμαστε βέβαιοι ότι οι τέσσερις άλλοι δεν θα κυρώσουν και ο ένας θα κυρώσει, επομένως δεν θα τεθεί σε ισχύ ποτέ, για να τεθεί σε ισχύ χρειάζεται πέντε. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε αυτό, γιατί αυτή ήταν η αρχική διαπραγμάτευση. Είμαστε βέβαιοι ότι άλλοι δεν θα κυρώσουν. Ένας κυρώνει, καλό είναι, αλλά πρέπει να το πούμε και στις άλλες αφρικανικές χώρες και κυρίως στη Δυτική Αφρική. Ένας ε, αρκεί να κυρώσει για να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά. Επιβεβαιώστε μου κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την Κένια, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και για άλλες αφρικανικές χώρες. Η Σάντρα, επιτρέψτε μου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εμεί έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν διαφορετικέ συνθήκε στι διάφορε χώρε. Η αναφορά στη Δυτική Αφρική δεν έχει ε, θέση εδώ, διότι είναι ε, τελείως διαφορετικές ενδιάμεσες συμφωνίες οι οποίες ε, ίσχυσαν εκεί. Η Κένια δεν έχει ενδιάμεση συμφωνία, επομένως είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου αυτό αυτός ο παραλληλισμός η συμβατότητα του ΠΟΕ και ε, το γεγονό ότι η ΜΑΡ δεν είναι συμβατή δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω. Εσείς μας βοηθήσετε να διευρύνουμε αυτό το θεματολόγιο, να έχουμε μια σχέση συμβατή ε, βάση ΠΟΕ με την Αφρική και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλό έδαφος γιατί αρχίζουμε να επιτυγχάνουμε ουσιαστικά να έχουμε μόνο μία χώρα υπό τη ΜΑΡ. Όλες οι άλλες χώρε θα έχουν μέσα τα οποία είναι συμβατά με το ΠΟΕ. Η ΣΑΝΤΕΚ θα είναι μια συμφωνία εταιρική σχέση η οποία θα είναι πλήρω συμβατή με βάση το ΠΟΕ. Η Τανζανία αυτή τη στιγμή πρέπει να το σκεφτεί, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποφασίσει να υπογράψει και να κυρώσει, θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία είναι πλήρω συμβατή. Ε, για το ΣΑΝΤΕΚ θέλω να τονίσω ότι θα υπάρχει κύρωση από όλες αυτές τις χώρες και είναι μια συμφωνία ε, εταιρική σχέσης. Ε, ε, θα απολαμβάνουν μια τέτοια συμφωνία. Μια τεχνική λεπτομέρεια, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Οι συμφωνίες αυτές έχουν ένα πολύ μακρύ πρόγραμμα εφαρμογής. Για παράδειγμα, ακόμα και το γεγονό ότι η Κάνα ή η ακτή του ελεφαντιστού ε, επιλέγουν να συμμετέχουν στην ενδιάμεση συμφωνία δεν θα δημιουργήσει στρεβλώσεις στην περιφέρεια, γιατί υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να αρχίσουν να ε, επηρεάζουν για να επηρεάσουν τη συμφωνία και θα περάσει μια δεκαετία μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Επομένω, σε δέκα χρόνια πιστεύουμε ότι θα την έχουμε κυρώσει τη συμφωνία. Είναι μια διαδικασία εν εξελίξη, δυναμική και σα παρακαλώ, σα ζητώ να, επιλεγού, ε, ε, να σεβαστούμε τι επιλογέ και να μην θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή είναι ένα πίνακα που πρέπει να εφαρμόζονται πράγματα. Δεν λειτουργεί έτσι η Ευρώπη. Κάθε χώρα γίνεται σεβαστή. Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση μια χώρα όπω η Κένια και για να είμαι ειλικρινή, έχουν την έγκριση των δικών του φορέων, τα δικούς τους θεσμούς, τους οποίους σεβόμαστε. Εάν υπάρχει μία όριμη απόφαση σε επίπεδο αρχηγού κράτου ότι πρέπει να υπογράψουν, η Κένια θα υπογράψει. Δεν χρειάζεται να ζητήσει την αδειά μα. Πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ του. Και ε, ε ήθελα απλώ να κάνω λίγο τη δασκάλα εδώ και να σας ζητήσω να μην κάνουμε συγκρίσεις με πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, ο τίτλος είναι Συμφωνία εταιρική Σχέσης, αλλά ε, ε, τα όσα ισχύουν ε, από κάτω είναι τελείως διαφορετικά. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένε ημερομηνίε για την υπογραφή και την κύρωση. Αναφερθήκατε στο Σεπτέμβριο, αλλά έχετε κάτι σαφέστερο να μας πείτε. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να υπογράψουμε. Θα θέλαμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία ήδη αύριο το πρωί, αν γινόταν. Αυτό είναι το σχέδιο μας. Δεν θα ε, επιστρέψω, δεν θέλω να επιστρέψω στην Κενέα χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία υπό τους όρους ε, της κύρωσης. Χθες ε, το βράδυ είπαμε ότι όταν θα διαλυόταν το κοινοβούλιο θα η συνεδρίαση του κοινοβουλίου την επομένη ήδη θα γινόταν τέλεια χρονική συγκυρία θα επιστρέψουν στις 2 Οκτωβρίου και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ως ημερομηνία λαμβάνουμε υπόψη και αυτό το στοιχείο δεν θέλουμε να χάσουμε την δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές ε, για μια μέρα όλοι και όλοι. Διότι πάρα πολλοί έχουν κάνει παραγγελίες ε, και θα μπορούσαν να υπάρχουν προβλήματα για επιχειρήσεις αν υπήρχαν κάποιες δυσχέρειες. Υπάρχει λοιπόν η δέσμευση και θα προχωρήσουμε σε σχέση με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επικυρώσουμε και να προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν ε, αυτή την πτυχή. Υπάρχει δέσμευση του, της κυβέρνησης της ε, Κένιας και θα προχωρήσουμε ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις αγορές. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ Εμπορίου. Ο Χέρμουτ Σόλτς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό και όλους τους ε, συναδέλφους για τη συμμετοχή για αυτή τη συζήτηση που έγινε και θα έπρεπε να μπορέσει να επιτευχθεί ή δυνατόν αύριο ήδη η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Από... Θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις και προτάσεις για όλες τις προτάσεις που έγιναν και να ευχαριστήσω για το αναβαθμισμένο περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων σε σχέση με την κοινοβουλευτική μας επιτροπή καθορίζοντας το πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, άλλες χώρες και σε σχέση με την προσέγγιση περιφέρειας προς περιφέρεια, region to region και πράγμα που και στην συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται ως πλαίσιο συνεργασίας με αυτές τις χώρες θα πρέπει να διαμορφώσουμε την άποψή μας σε σχέση με την ε, άποψή μας ε, για την εκύρωση αυτών των συμφωνιών και όλα αυτά θα πρέπει να αυξήσουν την ε, δυνατότητα κατανόησης για τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες, να κατανοήσουμε το πού βρισκόμαστε και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την οικονομική συνεργασία και σε σχέση με την συνεργασία περιφέρειας με περιφέρεια αλλά και σε σχέση ε, με, την πτυχή των επιμέρους χωρών δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε χώρα να προχωρήσει όπως εκείνη θεωρεί πιο εύθετο. Αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και για την χρονική παράμετρο των ε, ε, θεμάτων θα πρέπει να ε, βρεθεί ένα χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και ολοκληρώσαμε έτσι με αυτά τα θέματα για σήμερα το πρωί και το ίδιο συμβαίνει και με τις συζητήσεις ε, και για τη συζήτηση με τα θέματα της ε, Γκάνας. Μια και ο χρόνος πιέζει, θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή για να μας τα εκθέσει. <laughs> Είμαι σύντομος, είχαμε συζητήσει σχετικά και είχε συμπεριληφθεί το θέμα αυτό το 2008 και τώρα επιτέλους κύρωσε η Γκάνα καλύπτεται μέσω της ε, περιφερειακής συμφωνίας στην και ελπίζουμε ότι αυτή η εταιρική εμπορική σχέση θα μπορέσει να κυρωθεί και τον ε, Οκτώβριο να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως είναι μια εναλλακτική δύναμη, μια επιλογή αυτή που παραμένει ανοιχτή δεν είναι η ε, επιλογή που θα ε, θέλαμε να ισχύει κατά παρέκκληση, θα θέλαμε πράγματι να υπογράψει η Γκάνα. Είναι μια προσωρινή λύση αυτή η ε, διαδικασία όταν έχουμε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωσης και τα σχετικά. Καλύπτει ουσιαστικά η πτυχή αυτή την χωρίς δεσμούς, ε, δασμούς και τέλει πρόσβαση των αγαθών της στην αγορά που είναι το πιο σημαντικό και θα υπάρξει μια σταδιακή κλιμακούμενη απελευθέρωση των διαδικασιών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ε, προσωρινή διαδικασία και να δούμε και τη διάσταση της ε, περιφερειακής συμφωνίας εξίσου. Αλλά και πάλι αυτό αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας είναι η επιλογή την οποία έκανε η Γκάνα και έτσι θα ε, συνεχιστεί η διαδικασία. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε κατά την 1η Οκτωβρίου να έχουμε την κύρωση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να τεθεί σε λειτουργία η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από όλες τις συζητήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί, σε περίπτωση, στην περίπτωση της Γκάνας βλέπουμε ότι η άσκηση πιέσεων έχει τελικά ε, κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε σχέση με την απειλή που ε, σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον υπήρξε η ενδιάμεση συμφωνία που ε, ε, προχώρησε και μέσα σε ε, ξεχωριστό οικονομικό πλαίσιο και νομίζω είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον αν το λάβει κανείς αυτό υπόψη, σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση για την Κένια και την, ανατολική, ε, την κοινότητα των χωρών Ανατολικής Αφρικής σε σχέση με την πρόσβαση των προϊόντων τους για τις αγορές που την χάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης όσον αφορά τις επιμέρους προτιμήσεις ε, και δασμολογικές προτιμήσεις ε, ε, που ισχύουν εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό και αν δει κανείς το τι γίνεται με τις ε, συμφωνίες εμπορικής εταιρικής σχέσης καταλήγουμε σε μια ασύμετρη σχέση πραγμάτων που δεν είναι και η πιο εύθετη. Αν δει κανείς ε, την ενδιάμεση συμφωνία είναι πολύ διαφορετική από την Συμφωνία Εμπορικής Εταιρικής Σχέσης του 2014 και θα υπάρξουν και διαφορές ε, μέσα σε, σχέση με την ε, ε, ίδια την κοινότητα των χωρών αυτών και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προτεραιότητες που υπάρχουν σε σχέση με την συμβατότητα των όρων των συμφωνιών αυτών με τις διατάξεις του ΠΟΕ και όταν βλέπουμε ότι σε σχέση με τη συμφωνία του Κοτονού ή και την κοινωνία των πολιτών που ούτε μία φορά δεν αναφέρεται σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία ε, υπάρχει λοιπόν αντικατάσταση κάποιων ε, ε, ρητρών και η απουσία κάποιων ρητρών και θα έπρεπε πραγματικά αυτό να μας κάνει να ενδιαφερθούμε ιδιαίτερα και σε σχέση με το άμεσο μέλλον στην, η κατάσταση σε σχέση με την Ιγυρία δεν είναι η κύρια προτεραιότητα ε, που υπάρχει, το ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες σε σχέση με την Ιγυρία και όσον αφορά την κυβέρνηση της Νιγηρίας ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική και καταλήγουμε σε μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί παρόμοια με εκείνη της Γκάνας. Θα πρέπει λοιπόν να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι ο Υπουργός Εμπορίου της Κένιας παραβρέθηκε σήμερα εδώ και σε σχέση με την Ουγκάντα για τα θέματα επικύρωσης ε, για την ε, αύξηση των ε, εξαγωγών της Ουγκάντα και σε σχέση με την την άποψη που εκφράζεται ότι εδώ υπάρχουν ισομερείς σχέσεις, ισόρροπες σχέσεις, όταν βλέπουμε να ασκούνται πιέσεις ε, και να επισύονται απειλές ε, ε, σε σχέση με κάποιες χώρες και για την τελευταία παρατήρηση το κυριότερο θέμα εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ότι οι ενδιάμεσες συμφωνίες που δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει κανείς παραπέρα ίσως να υπονομεύουν κιόλας και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Πρέπει να προωθούμε την οικονομική συνεργασία και εμπορική συνεργασία μεταξύ ομόρων χωρών και μέσα στο πλαίσιο αυτό να δράσουμε. Πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα λοιπόν και να μην υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια όσον αφορά τα, τις ε, ε, γειτονικές χώρες. Πρέπει λοιπόν πραγματικά εδώ σκηνοβούλιο να ε, δράσουμε βλέποντας την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντς, ε, ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομος πρόεδρε σε σχέση με την ε, εταιρική αυτή εμπορική σχέση θα προτιμούσαμε να υπήρχε μια περιφερειακή συμφωνία κοινοτήτων χωρών ε, έχω και κάποιες ερωτήσεις ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσταση στην Ιγυρία συγκεκριμένα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσε να δώσει. Γιατί δεν ήταν σε θέση να υπογράψει η Νιγηρία αυτή τη συμφωνία. Γιατί η πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση είτε δεν ήταν σε θέση είτε δεν επιθυμούσε να το πράξει. Τι θα γίνει τώρα. Θα υπογραφεί ή δεν θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία και πώς θα αντιμετωπιστεί και θα επιλύει αυτό το πρόβλημα. Και τι κάνετε εσείς, ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε για να αντιμετωπιστεί και να διευθετηθεί αυτό το πρόβλημα. Και σε σχέση φυσικά και με την Γκάνα να δούμε το τι θα γίνει σε σχέση με τα θέματα ενδιάμεσων συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σόλτσε δεν είναι εδώ και ο δυσίγητης μας, αλλά θέλω να κάνω μια περαιτέρω παρατήρηση που δεν ακούστηκε. Δεν αντιλαμβάνομαι απολύτως γιατί δεν έγινε... Ε, διότι η ενδιάμεση συμφωνία έχει τελείω διαφορετικέ ε, δασμολογικέ γραμμέ σε σχέση με αυτέ οι οποίε ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση στη Συμφωνία τελική Σχέση. Αυτό σημαίνει ότι το περιφερειακό πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε το 2007. Και επομένως θεωρώ ότι η κύρωση και η προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας θέτει εν κινδύνο την περιφερειακή συνεργασία. Γιατί να μην εφαρμόζεται για την Κάνα η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για την Γένεια. Να παραμείνουν δηλαδή στη ΜΑΡ. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, η ακτή του ελεφαντιστού έχει μία έκπτωση δασμών και τώρα πρέπει να αλλάξουν την ε, ε, γραμμή, είναι προς το βαρύς, ενώ στην Κάρνα είναι πιστοβαρής. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω και πώς να το πω στα αγγλικά, ουσιαστικά σοκάρουμε την περιφερειακή συνεργασία. Και τρίτο, αυτό είναι πολιτικής φύσεως. Αν δείτε τις ε, ε, διάφορες χώρες ε, της ECOWAS, της Δυτικής Αφρικής, δείτε τι γίνεται στο Μαλί. οι πιέσεις μας πραγματικά οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας και συμφωνούν και οι πολίτες διότι υπάρχει μια πολύ περίπλοκη πολιτική και κοινωνική κατάσταση, την οποία εκμεταλλεύονται άλλε δυνάμει για του δικού του τους στόχου. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά όταν εμεί αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στην ε, ε, πυρηνική βιομηχανία της Γαλλίας και την παρουσία της στο Μαλί. Ε, και τι γίνεται με τις διάφορες πιέσεις από ισλαμικές ομάδες και το καθεξής υπησερχόμαστε ουσιαστικά στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω όταν ε, ε, εξετάζουμε μόνο τις εμπορικές πτυχές και δεν εξετάζουμε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σόλτς για αυτή την πολύ τεχνική ερώτηση. Ε, ε, είπατε διαφορετικές ε, δασμολογικές γραμμές. όχι. Στην ουσία προσφέρουμε τα ίδια πράγματα, κάποιες περιφερειακές αλλαγές, στις παρυφές αν θέλετε, η αρχή της εφαρμογές είναι πανομοιότυπη με ε, τη Συμφωνία εταιρική ε, Σχέσης που έχουμε για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Υπάρχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα βέβαια, αλλά αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι υπάρχει διαφορετική ε, ονοματολογία. Έχουμε τη συμφωνία του 2008 και πρέπει αυτό να το μεταφράσουμε στα, τη συμφωνία του 2012 συζητήθηκε και αυτό το τεχνικό ζήτημα με τον αρμόδιο υπουργό, το Χάνα Τέτε, αλλά είναι απλά τεχνικό ζήτημα. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Θα ήθελα τώρα να πω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Γκάνα είναι μια οικονομία που είναι διαφοροποιημένη. Έχει προϊόντα προστιθέμενης αξίας, έχει ε, στοιχεία τα οποία ε, πρέπει να εξάγονται με προτιμησιακό καθεστώς εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτά είναι καλά νέα για μας και παρεπιπτόντως η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ε, προϊόντων προστιθέμενες αξίας από την Αφρική, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Νιγηρία εξάγει πετρέλαιο. Επομένως, δεν μπορείτε στην ουσία να πείτε ότι επιλέγουμε τις σχέσεις μας. Πρόκειται για κυρίαρχη απόφαση των διαφόρων χωρών και μια χώρα που έχει πολύ περιορισμένη διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή δεν θα την πιέσουμε κατεπηγόντως ε, για να ε, συνάψει μια συμφωνία για προτιμησιακό καθεστώς. Σα το λέω για παράδειγμα ότι για την Ιγυρία υπάρχει ολόκληρη συζήτηση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές άλλες προτεραιότητες και η κυβέρνηση δεσμεύεται πλήρως ε, για να προωθήσει τις συζητήσεις. Ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου ε, έρχεται σε επαφή μαζί μας τακτικά και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνουμε σε συνεδριάσεις που ε, διοργανώνουν. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία που ξεκινούν αυτοί εσωτερικά ε, και χαιρόμαστε γι' αυτό γιατί οι Νιγηριανοί ε, φροντίζουν για το μέλλον τους και καταλαούν ότι το να εξαρτώνται από ένα αγαθό και μόνο και μάλιστα το πετρέλαιο με όλες αυτές τις διακυμάνσεις και τις αστάθειες που έχει φυσικά θα δημιουργήσει προβλήματα γι' αυτό προσπαθούν να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους. Η Γκάνα ήταν ιδιαίτερα υπομονετική με την υπόλοιπη περιοχή διότι η Γκάνα περιμένει από το 2007, μην σας πω και από το 2006, διότι το 2006 αντιλήφθηκαν ότι δεν θα υπάρχει ακόμα περιφερειακή συμφωνία, επομένως επέλεξαν την ενδιάμεση συμφωνία και ε, τελικά περίμεναν για τη συμφωνία, για την υπογραφή και περίμεναν και για την κύρωση μέχρι τώρα. Αλλά τώρα θέλουν να μην απειλούνται συνεχώς οι επενδυτές τους ε, ε, με πάυση του καθεστώτος. Εμείς δεσμευόμαστε να καταλήξουμε στην Περιφερειακή Συμφωνία, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να έχουμε Περιφερειακή Συμφωνία, όπως εξήγησε και ο εισηγητής, είναι μια καλύτερη συμφωνία, Περιφερειακή Συμφωνία, ιδίω όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, ε, κανόνες προέλευσης. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε Περιφερειακή Συμφωνία. Επιμένω λοιπόν ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία θα αναπτυχθεί σταδιακά και φυσικά η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ε, δεδομένων και των όσων είχαμε στην αρχή, ε, δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις στην περιοχή και ε, τα πάντα θα μας οδηγήσουν σε μια περιφερειακή συμφωνία. Ελπίζω λοιπόν να καθησύχασα λίγο τους φόβους σας. Η Γκάνα έχει επιλέξει να ακολουθήσει ένα μέσο το οποίο ήδη είχε επιλέξει το 2007 γιατί περιμένει να κινηθεί η υπόλοιπη περιοχή αλλά ακόμα δεν έχει κινηθεί. Ε, παρεπιπτόντως να σας πω ότι έχω βάσιμες ελπίδες ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, διότι το 2007 δεν υπήρχε ε, ένας κοινό εξωτερικός δασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Συμφωνία ECOWAS. Υπάρχει πραγματικά ένας κοινό εξωτερικός δασμός που πραγματικά σημαίνει ότι θα προχωρήσουν στην Περιφερειακή Συμφωνία πολύ πιο εύκολα. Δεν είχαμε κατά αντίστοιχο στο παρελθόν. Μπορεί να είχαμε στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν υπήρχε. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινό εξωτερικός δασμός και ε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα η Νιγηρία θα ε, προχωρήσει και αυτή στην ε, Συμφωνία εταιρική σχέση. Ευχαριστώ κύριο Φιέλνερ. Συμφωνώ με την Τζουτ για τις αδυναμίες της συμφωνίας, αλλά έτσι είναι στον κόσμο και στη συμφωνία αυτή. Εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε ένα σωρό πράγματα που λείπουν από τη συμφωνία. Η προσωρινή Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει κάποια ασφάλεια στους εταίρους και από τους εταίρους. Καταλαβαίνω ότι η Γκάνα θέλει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον λύγει το ΜΑΡ. Όταν μιλάμε για πυλές, ότι πιέζουμε, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί συμφωνήσαμε ότι το ΜΑΡ σταματάει κάποια στιγμή. Το συμφωνήσαμε, η πλειοψηφία του σώματος. Και η δικιά σας ε, η ομάδα διαπραγματεύτηκα με τους συναδέρφους σας. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι τελειώνει το ΜΑΡ και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου ρεαλιστικά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μεμονωμένα την κάθε χώρα. Συμβαίνει αυτό που εμείς αποφασίσαμε ότι θα συμβεί. Και ακόμα και αν ακούγεται ότι εμείς πιέζουμε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την άποψη. Ακριβώς η Γκάνα θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη λύση, γι' αυτό ακριβώς και την φτιάξαμε και είμαστε εμείς που συμφωνήσαμε ότι το ΜΑΡ θα σταματήσει κάποια στιγμή. Έχει ημερομηνία λήξη. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά θα συνεχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα, αν μας έρθει έτοιμα από το Συμβούλιο. Καλώς. Τώρα έτσι η δημόσια συνεδρίαση έληξε και αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών σε λίγο.